Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία της οποία είχε διακοπή. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο υπαριθμών 8 ακρόαση της Επιτροπής για τον έλεγχο του προϋπολογισμού για το EFSF και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας καθώς και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ESM. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που στη σημερινή μας συνεδρίαση έχουμε διακεκριμένους ομιλητές για το θέμα αυτό αριστερά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλώς ήρθατε κύριε Καλδέρα. Εκτιμούμε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήρθατε εδώ γιατί είναι μια ε, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου αντιπροσωπεία υπό την προεδρία του κυρίου Λαμασούρ, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης το ελεγκτικό συνέδριο του Λουξεμβούργου και εκτιμούμε πάρα πολύ το γεγονό ότι θα εδώ, να, αποφασίσετε να παραστείτε εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για να μιλήσουμε για το εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα, πώς μπορεί να υποβάλει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σε έναν δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών μελών και ενδεχομένως να επιφέρει βελτιώσεις. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ιβάνοφα η οποία είναι η συγγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει επευθερωθεί το θέμα αυτό. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, όταν οι συντονιστές στην συνεδρίασή τους στις 26 Ιανουαρίου 2012 αποφάσισαν να διοργανώσουν την τη σημερινή ακρόαση. Υπήρχε η ελπίδα ότι σήμερα είτε θα έχουμε επαρκείς πληροφορίες εν σχέση με, τον... με την έκταση, τον τρόπο λειτουργίας ε, των διαφόρων ε, τμήματων των οργάνων αυτών ή ότι θα ε, ή θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την αναγκαιότητα όλων αυτών των μηχανισμών. Αλλά δυστυχώς δεν είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επισέλθουμε περισσότερο στα θέματα αυτά γιατί πρέπει να το κάνουμε. Θα ήθελα να αναφέρω μια γνωμοδότηση οικονομολόγων ε, για παράδειγμα τον επικεφαλής του, της Γερμανικής, ε, του Γερμανικού Ταμιευτηρίου, ο οποίος διαπιστώνει ότι οι λόγοι της ε, διαρθρωτικής ε, κρίσης δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστούν στο επίπεδο των χωρών μελών, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική ανάπτυξης ε, που να δώσει δυνατότητα στις χώρες μέλη να επανέλθουν στους κόλπους Οικονομικής και Νομισματικής Ενότητας. Τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο ε, δεσμεύονται στο έργο της εξέτησης μεν κομισιόν να αναλάβει ένα κεταμένο εποπτικό έλεγχο, το δε Συμβούλιο να δεσμεύεται προς τις χώρες μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν έχει ούτε εποπτικό ρόλο, ούτε ρόλο ελέγχου. Και αυτό ισχύει τόσο για το EFSF τόσο, όσο και για το ESM. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα, υπάρχει ένα χάσμα όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων που κατά την άποψή μου κατά κανένα τρόπο δεν, έχει γίνει κατανοητή από τους ε, πολίτες και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να αρθεί αυτό το χάσμα, να απαλληφθεί αυτό το χάσμα. Και διότι πρόκειται για μια βασική αρχή ε, της, ε, των δημοκρατικών συστημάτων να μεριμνούν ούτως ώστε οι δαπάνες των δημοσίων κονδυλίων και ε, να μην ε, είναι δυνατόν να εκτίθενται σε κινδύνους χωρίς να υπάρχει, να ασκείται ένας δημοκρατικός έλεγχος. Αλλά όλες αυτές οι διαπιστώσεις επισημαίνουν ότι παρόλα αυτά ε, θα πρέπει εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επεξεργαστούμε περισσότερο το θέμα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των μηχανισμών. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και ειδικού που θα διευκρινίσουν αυτές τις ε, πτυχές. Ήδη για το τον προηγούμενο χρόνο και για το 2009 οι βουλευτές της Επιτροπής μας τόνισαν τη σημαντικότητα των μηχανισμών ελέγχων των διαφόρων ε, μηχανισμών ε, διάσωσης. Σε σχέση με το ESM, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ήθελε να έχει μία ε, ενδεδειγμένη ε, λογοδοσία ούτως ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της βάσης των δεδομένων η έκθεση απαλλαγή τη Επιτροπής, η οποία έγινε, εγκρίθηκε από την Επιτροπή τέλη Μαρτίου, επαναλαμβάνει αυτά τα αιτήματα και διευκρινίζει ότι το καταστατικό του ESM, που προ το παρόν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευση εξ μέρου των χωρών μελών, ε, θα πρέπει να προβλέψει ε, τέτοιες διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσία. Αυτή ε, τη στιγμή θα, στο πλαίσιο αυτής της ακρόασης θα συζητήσουμε τον τρόπο που ασκείται αυτός ο δημοκρατικός έλεγχος. Ε, επιτρέψατε μου να σας παρουσιάσω τους πέντε ομιλητές που καλέσαμε. Καταρχή έχουμε τον Ρόλαν Ζανκάρ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την μελέτη του για την αξιοπιστία του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το EFSM και το ESM και την ε, σημασία του ελέγχου του προπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια έχουμε την Κάλιν Ανέφ, τη Γενική Γραμματέα του EFSF και στη συνέχεια το Μάρκο Μπούτι, Γενικό Διευθυντή ε, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών ε, Υποθέσεων. Στη συνέχεια έχουμε την, θα έχουμε την ομιλία του κυρίου Βίκτορ Καλδέρα, ε, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Χόρστ Ερμπ, ο οποίος είναι ελεγκτής ε, διευθυντής και μέλος του Bundesrechnungshof, του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Κέσ Βέντρικ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μάλλον είχε προγραμματιστεί ο κύριος Κέσ Βέντρικ, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εδώ και θα αντικαταστεί από τον κύριο Γιάννε Βάντες ο οποίος είναι ειδικευμένο στα θέματα αυτά. Οι εκπρόσωποι των ελεγκτικών συνεδρίων θα μιλήσουν από τη σκοπιά των ελεγκτικών συνεδρίων των χωρών αυτών και θα μιλήσουν για, το, για την υποχρέωση λογοδοσίας και το πώς τα ελεγκτικά συνέδρια ενέχονται στο ρόλο αυτό του ελέγχου των μηχανισμών ε, διάσωσης. Ε, έχουμε τρία τμήματα σε αυτή τη συνεδρίαση ε, θα μιλήσουν καταρχήν οι μελητές και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Και ε, θα μιλήσουμε με τη σειρά που σας ε, παρουσίασα. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που η ακρόασή μας έτυχε ε, τη χάνει τόσο μεγάλο ενδιαφέροντο ε, μεταξύ των προσκεκλημένων μας και όλα αυτά τα χρωστούμε μεταξύ άλλων στην πρωτοβολία της Αντιπροέδρου μας ε, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και στην εισηγήτριά μας, κυρία Ελιάνα Ιβάνοβα, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και μας υπέβαλε μια πολύ καλή έκθεση. Παρακαλώ την κυρία Ιβάνοβα να μας κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση στο θέμα μας. Ευχαριστώ συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού οργανώνει σήμερα αυτή την ακρόαση. Περνάμε δύσκολε και ενδιαφέρουσε εποχέ. Το δημόσιο χρέο έφτασε αφόρητα επίπεδα σε κάποια κράτη-μέλη και η παρέμβαση Ευρωπαϊκή Ενώσεω ήταν υποχρεωτική για να διασώσει την Ευρωζώνη. Πέρσι εδώ στο Κοινοβούλιο συμφωνήσαμε επί τη δέσμη των έξι μέτρων για την ενίσχυση τη οικονομική διακυβερνήσεω στην Ευρωζώνη. Όμως αυτή η δέσμη μέτρων θα δώσει αποτελέσματα μέσω μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα η Ευρώπη χρειαζόταν κατεπηγόντως μέσα για οικονομική βοήθεια για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Και σχετικά με αυτό, θα ήθελα να πω ότι το 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει δύο προσωρινά μέσα για την οικονομική βοήθεια προ τα κράτη-μέλη, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Οικονομική Σταθερότητα και το Ευρωπαϊκό Μέσο Λοιπόν, ο μηχανισμό σταθερότητα θα, θα αντικαταστήσει αυτά τα δύο μέσα και θα λειτουργήσει από φέτο τον Ιούλιο. Ακόμα και αν οι μηχανισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή να παράσχουν βοήθεια στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή που απειλούνται από σοβαρέ οικονομικέ δυσκολίε, είναι διαφορετικά σε δομή τρόπου χρηματοδότηση και συστήματα ελέγχου προϋπολογισμού. Αυτή η ακρόαση έχει στο στόχο μας ενημερώσει για την όλη κατάσταση, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν σήμερα για το ESFF και για το e FSM και να γίνει μια αξιολόγηση της νέας συνθήκης ESM για σταθερότητα όσον αφορά τον έλεγχο. Ε, χαίρομαι που έχουμε διάφορους ενδιαφερομένους που εκπροσωπούνται εδώ από, το, από τους ίδιους μηχανισμούς σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς και σας καλωσορίζω όλους τι ακριβώς θα συζητήσουμε σήμερα όσον αφορά τα τρία αυτά χρηματοπιστωτικά μέσα. Το FSM δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να δανειστεί πάνω μέχρι 60 δις ευρώ από τι αγορέ κεφαλαίων και να τα δώσει στα κράτη-μέλη, τα δανεί στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Τα δάνεια υπό το EFSM στηρίζονται από κοινοτικά χρήματα, τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και είναι φυσικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει τη δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του, της προπολογισμού και απαλλαγή Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει αυτό λόγο να παίξει σαν εξωτερικό ελεγκτής του FSM και μπορεί να διενεργήσει ελέγχου οικονομικών επιδόσεων όσον αφορά διανοδότηση και διανοληψία, πλευρά τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το FSM είναι ειδικό μέσο που, ε, στο οποίο συμμετέχουν τα κράτη-μέλη, έχουν δεσμευτεί. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αναμειγνύεται καθόλου στον έλεγχο του τρόπου λειτουργία του και το FSF e δεν συμπεριλαμβάνει δικαιώματα ελέγχου από πλευράς των ελεκτικών φορέων και επίση δεν προβλέπεται εξωτερικό έλεγχο. Το ESM με τη σειρά του θα είναι ένα διεθνή φορέα που δημιουργείται από τη Συνήθεια Ευρωπαϊκή Ενώσεω, θα χρηματοδοτείται μέσω ενός κεφαλαίου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ και δάνεια μέχρι 680 δισεκατομμύρια ευρώ. Ασχολείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον έλεγχο ε, του ESM ε, και επίσης και οι ανώτατοι ελεγκτικοί φορείς ασχολούνται με αυτό το θέμα, προβληματίζονται διότι δεν καλείται επαρκώς το θέμα από πλευρά της ε, συνθήκης για τον εξωτερικό έλεγχο. Ο εξωτερικός δημόσιος έλεγχος του ESM θα διενεργείται από το ελεγκτικό συνέδριο όπου από ελεγκτικό συνέδριο και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο συμμετέχει στο φορέα αυτόν μαζί με τα δύο μέλη που εναλλακτικά θα ορίζονται που θα εκπροσωπούν τους ανώτατους ελεγκτικούς χωρίς. Πέρσι είχα διοριστεί εισηγήτρια για μια ειδική μελέτη όσον αφορά την, ε, το EFSM και το ESM σχετικά με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και πώς μπορεί να αναμειγνύεται στον έλεγχο τον οικονομικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Σήμερα στο πρώτο πάνελ θα παρουσιαστεί αυτή η μελέτη και θα εστιαστεί επί της επαρκείας του FSM και το ESM, σχετικέ διατάξεις που αφορούν τους ελέγχους. Επίσης θα αναφερθούμε σημαντικά θέματα όπως είναι οι δέουσες διευθετήσεις για τους δημόσιους εξωτερικούς ελέγχους, πλήρη διαφάνεια για τον μόνιμο μηχανισμό της κρίσης, αξιοπιστία στοιχείων, στατιστικών, ευθύνες, ενημέρωση πλευράς εμπλεκομένων φορέων και βεβαίως ο πολιτικό έλεγχο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Σημαντική πτυχή για την οποία είμαι ευγνώμων που συμπεριελήφθη στην ανάλυση είναι το μέσο για τον ισολογισμό των πληρωμών. Είναι ένα άλλο μέσο για να υποστηρίξει τα κράτη που δεν είναι στην Ευρωζώνη και αντιμετωπίζουν σοβαρέ οικονομικέ δυσκολίε διότι αυτό το μέσο προσθέτει άλλα 50 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στο ευρωπαϊκό προπολογισμό, διότι τα δάνεια στηρίζονται εκ νέου από κοινοτικού πόρου και καλωσορίζω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που εξέφρασε προθέσει να συμπεριλάβει μια αναθεώρηση του μέσου για την εξυπηρέτηση των ισολογισμών στο πρόγραμμα ελέγχου για το 2012. Το δεύτερο πάνελ, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, θα εξετάσει ενδελεχέστερα το θέμα του δημοσίου ελέγχου των τριών μέσων, Ποιο είναι ο ρόλο του διαχειριστού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, και στο τρίτο πάνελ θα συζητήσουμε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πτυχές όσον αφορά τους ενέχους και στροπτικές προσφέροντες, συνοψίζοντας έχουμε 60 δισεκατομμύρια από το EFSM, συν 50 δις από το μέσο των ισοζύγιο πληρωμών, 110 δις ευρώ όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό που θα τα καταβάλει, ε, που θα είναι όλες πληρωμές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που δεν έχουμε αμφισβητήσει, δεν έχουμε εξετάσει σε το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τέσσερα ακρόασης ελπίζω να έχουμε σαφείς απαντήσεις για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Ήρθε η ώρα να τεθούν αυτά τα ζητήματα, το χρωστούμε στους πολίτες, στους φορολογούμενους Ευρωπαϊκής Ενώσεως και προσβλέπω σε μια καρποφόρα συζήτηση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, dear... Ευχαριστώ πολύ αγαπητή συνάδελφε Ιβάνοβα για αυτή την εισαγωγή στο σημαντικότατο θέμα. Και τώρα καλό να έρθει εδώ ο κ. Σονκάρα από την PricewaterhouseCooper. Καλώς ήρθατε. Να έρθετε να κάνετε την παρουσίασή σας, τη μελέτη, να μας παρουσιάσετε τη μελέτη που αναλάβατε. Μεγάλη χαρά για μας που ήρθατε εδώ. Και ήρθατε να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα. Καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο λοιπόν αγαπητέ κυρία. Uh, uh, κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχει σήμερα η PricewaterhouseCoopers να παρουσιάσει τα βασικά της πορίσματα κατόπιν διεξαγωγής μελέτης Ονομάζομαι Ζανκάρ και εργάζομαι στην ε, PwC του Βελγίου. Έχω άλλους δύο-τρεις συναδέλφους εδώ με στην αίθουσα που έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για την προετοιμασία της έκθεσης. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν και έχετε λάβει όλοι ένα αντίτυπο της μελέτης ε, προδημοσίευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το disclaimer της μελέτης γιατί σε σχέση κυρίως με το ESM ακόμη προετοιμάζονται πάρα πολλά έγγραφα και άρα είναι διαβαθμισμένα. Βασιστήκαμε λοιπόν για την διεξαγωγή της μελέτης σε έγγραφα που είναι διαθέσιμα στο κοινό. Θα ακούσουμε και τις παρατηρήσεις σας και αν χρειαστεί θα προσαρμόσουμε αναλόγως ε, την ε, έκθεσή μας. Ποιος ήταν ο στόχος λοιπόν της μελέτης. Όπως ανέφερε η κυρία Ιβάνοβα, Μα ζητήθηκε να εξετάσουμε την ε, λειτουργία δύο μηχανισμών για την διευθέτηση κρίσεων. Πρώτον το EFSM, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δημοσιονομικής Σταθερότητας, ο οποίος ε, ιδρύθηκε το 2010. Όπως ε, εξήγησε η κυρία Ιβάνοβα, χάρη σε αυτό το μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να δανειστεί στις κέφαλαια αγορές ούτως ώστε στη συνέχεια να δανείσει αυτά τα κεφάλαια στα ε, κράτη-μέλη που ανήκουν στην Ευρωζώνη και αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η άλλη οντότητα, ο άλλος μηχανισμός που μελετήσαμε είναι ο ESM, είναι ένας νέος μηχανισμός, ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας ε, η σχετική συμφωνία για τη θέσπιση του εγκρίθηκε προσφάτως και ως νομική οντότητα θα έλεγα ότι συνιστά ένα διακρατικό οργανισμό με πρικοδότηση 80 δις. Όπως αναφέρατε, η δανειοδοτική δραστηριότητα θα υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη και άρα δεν επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίσαμε τη μελέτη μας λοιπόν για το EFSM και ESM σε πέντε διαφορετικές ε, θεματικές ε, ενότητες. Ε, η ρόλη των δύο μηχανισμών και οι ευθύνε που αυτοί συνεπάγονται, η επάρκεια του ελέγχου του προπολογισμού, ρυθμίσεις για εξωτερικό έλεγχο, αξιοπιστία δεδομένων και στατιστικών, καθώς και δημοκρατικός έλεγχος. Βασιστήκαμε σε αυτά τα έγγραφα που προανέφερα για τη διεξαγωγή της μελέτης. Κάναμε επίσης διάφορες συνεντεύξεις. Στο παράρτημα 3, αν θυμάμαι καλά, της έκθεσής μας βρίσκεται όλους όσους ε, ε, μετήχαν στην μελέτη και έδωσαν συνέντευξη. Έχουμε και μία ε, σύνοψη. Μετά από την σύνοψη ακολουθούν οι συστάσεις και στη συνέχεια τα πιο λεπτομερή πορίσματα. Θα ήθελα τώρα εντάχει να εξετάσω μαζί σας ε, την ε, σύνοψη. Πρώτον, ε, όπως σας είπα, ο ρόλος και η ευθύνη κάθε μηχανισμού. Στις σελίδες 11 και 12 της έκθεσής μας βλέπετε αυτά τα στοιχεία. Σε σχέση με το EFSM, όπως σωστά είπε η κυρία Ιβάνοβα, η κατάσταση, το καθεστώς ε, που ισχύει προσωμιάζει άλλα προγράμματα δημοσιονομικής αρρωγής, παραδείγματος χάρη ο μηχανισμός βασίζεται στο ισοζύγιο πληρωμών, ε, ή ε, ο μηχανισμός της μακροοικονομικής αρρωγής, MFA. Είναι συγκρίσιμα τα καθεστώτα σε περιπτώσεις φυσικά όπου συντρέχει λόγος για χορήγηση επίγουσας ε, οικονομικής βοήθειας. Σε σχέση με τη λειτουργία του EFSM υπάρχει ευρύτατη τεκμηρίωση διαθέσιμη και κοινοποιείται ε, σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και το Κοινοβούλιο. Χορήγηση δανείων λοιπόν προς το Συμβούλιο και ενημέρωση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε απόφαση δανειοδότησης. Η κατάσταση για το ESM διαφέρει λόγω της νομικής του φύσης. Πρόκειται για μια διακρατική ε, οντότητα, διακρατική θεσμική αρχή και δεν εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. μελετήσαμε και τη συνθήκη και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για κάποιες επιτυχές οι διατάξει της συνθήκης ε, συνάδουν με τις απαιτήσεις του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφέρομαι ε, στην σχετική έκθεση που εξέδωσε το Κοινοβούλιο Κατά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ε, κάποιες ε, οντότητες, κάποιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκονται, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει άμεση και έμεση εμπλοκή λοιπόν διαφόρων φορέων Ε, στα πλαίσια του ESM η διακυβέρνηση μοιάζει με τη διακυβέρνηση άλλων διεθνών φορέων όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το EFSF, Η διακυβέρνηση λοιπόν έχει ευθυγραμμιστεί με τη διακυβέρνηση άλλων διεθνών φορέων θα ήθελα να ευσύσω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Όπως σας είπα και νωρίτερα, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ε, τα bylaws, ε, δηλαδή τις παράγωγες διατάξεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Ε, ως προς τη λειτουργία του ESM Υφίστανται επίση ε, διαδικασίες ε, που ακόμη δεν έχουν ε, προσδιοριστεί τελεσίδικα, παραδείγματο χάρη η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εσωτερικό έλεγχο, το, ελεγκτικό, το εσωτερικό ελεγκτικό συμβούλιο, και η σχέση με τα SAIs, δηλαδή τα, τις ανώτατες ελεγκτικές αρχές. Δεύτερον, έλεγχος ε, του προϋπολογισμού. Η FSM πρώτα απ' όλα. Η δανειοληψία, δανειοδοσία βάσει αυτού του μηχανισμού ε, καταγράφονται στους λογαριασμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρα ελέγχονται από τις πολιτικές αρχές μέσω της έγκρισης ε, του προπολογισμού και της χορήγησης απαλλαγής. Καθότι αυτό συνιστά ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, υπάρχει το μηχανισμός ε, σε ελέγχους και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Κοινοβούλιο έχει στη διάθεσή του πάρα πολλές πληροφορίες για τη λειτουργία του EFSM, μεταξύ των οποίων και οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Ως προς το ESM και λόγω της νομικής του φύσης, η διακυβέρνηση, αιτήσει, λογαριασμοί εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αιτήσει, αυτοί οι λογαριασμοί θα είναι διαθέσιμοι για ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια, τις Ανώτατες Ελεγκτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ελέγχονται οι λογαριασμοί επίσης από εσωτερικό ελεγκτή και θα πιστοποιούνται από εξωτερικό ελεγκτή. για την ε, παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων ε, θα έχει την ευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προσδιορίζει τις διαδικασίες για την ε, δημοσιονομική διαχείριση και τη διαχείριση κινδύνου. Για τη διαχείριση κινδύνου προτείνουμε ως προς το ESM να ακολουθηθεί η αρχή της διαχείρισης κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής αρχής τραπεζών. Ε, το, στο EFSM, όπως είπαμε, προβλέπονται οι οικονομικοί έλεγχοι από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για τους ετήσιους λογαριασμούς. Επίσης, μπορούν να κάνουν ελέγχους ε, συμμόρφωσης και απόδοσης. Ο κύριος Καλντέιρα στη συνέχεια ε, πιστεύω θα μας εξηγήσει το έργο του ελεκτικού συνεδρίου ως προς το EFSM. Για το ESM οι ελεγκτικές ε, δραστηριότητες εποπτεύονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι μια ελεγκτική επιτροπή που θα εποπτεύει η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου καθώς και την υπηρεσία εξωτερικού ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παραδείγματο χαρή, εμέσω ε, θα ε, παρεμβαίνουν στο ESM. Επίση, ε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει τι δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα αυτό, δηλαδή ω προ τη ESM. Αν προκύψουν διοικητικά και σε δαπάνες ε, στην όλη διαδικασία θα ελέγχονται επίσης ε, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τέταρτη θεματική ενότητα που κληθήκαμε να εξετάσουμε τώρα. Αξιοπιστία των δεδομένων και των στατιστικών στοιχείων. Για το EFSM η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί δεδομένα που προέρχονται αφενός από την Eurostat, αφετέρου από τα κράτη-μέλη. Στο παρελθόν ε, δημιουργήθηκαν προβλήματα σε σχέση με τα δεδομένα, αλλά τρέχουν αυτή τη στιγμή ε, μεγάλου εύρους προγράμματα με στόχο την αναβάθμιση των στατιστικών στοιχείων, παραδείγματος χάρη επιτόπου έλεγχη, καθώς και ε, ενοποίηση ε, διαφόρων ε, βάσεων κόμβων προσκόμισης στοιχείων από πλευράς των κρατών μελών. Ο στόχο είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων. Τι συμβαίνει τώρα στα πλαίσια του ESM. Ουσιαστικά μιλάμε για τα ίδια δεδομένα που προέρχονται από την Eurostat και από τα κράτη-μέλη. Άρα δεν έχω να κάνω κάποια ξεχωριστή παρατήρηση. Ισχύουν αυτά που σας είπα για το EFSM. Για τα αμυγό οικονομικά στοιχεία του ESM τώρα, οι λογαριασμοί και άλλα τέτοια οικονομικά στοιχεία. Όλα αυτά θα είναι συνάρτηση του αποτελέσματο ε, του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου καθώ και τη διαδικασία διαχείριση κινδύνου. Τελευταία θεματική ενότητα που εξετάσαμε είναι ο δημοκρατικός έλεγχος για το EFSM, όπως σας είπα, και το ίδιο ισχύει για το μηχανισμό ισοζυγίου πληρωμών και το μηχανισμό μακροοικονομικής ε, βοήθειας, ε, MFA. Ε, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, έχουμε τα μνημόνια συνεννόησης, τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωμοδοτήσεις και ελέγχους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Επίσης ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει στοιχεία ε, επ' αυτών και δύναται να ε, ασκήσει αυτόν τον δημοκρατικό έλεγχο. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Κάποια στιγμή θα τερματιστεί η λειτουργία του EFSM και τα δάνεια που θα συνεχίσουν να υπάρχουν παρόλα αυτά, παρά την πάυση λειτουργία του μηχανισμού, είναι το θέμα που μας απασχολεί, γιατί θα πρέπει να παρακολουθούμε την όλη διαδικασία σε σχέση με το ESM. Ε, υπάρχει δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά όχι μόνο, Τα Εθνικά Κοινοβούλια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα λαμβάνουν τακτικά ενημέρωση για τους ετήσιους ε, λογαριασμούς του ESM. Και άρα βάσει των αρχών διακοινοβουλευτικής συνεργασίας ανάμεσα αφενός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ε, προκύψει κάποιο είδους έλεγχος. Το θέμα προσυζήτηση είναι... Α, ναι οι οι λογαριασμοί του ESM που θα προετοιμάζει το Διοικητικό Συμβούλιο θα κοινοποιούνται στα, ευρωπαϊκά, στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως είπαμε, αλλά τίθεται το ζήτημα θα πρέπει να διαβιβάζονται αυτά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδού, σαν δρές γραμμές, ε, η, τα πορίσματα ε, της έκθεσής μας και ε, είμαι στη διάθεσή σας αν υπάρχουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ζανκάρ για την παρουσίασή σας. Ε, ουσιαστικά ορίζεται ένα πλαίσιο με την παρουσίασή σας ε, και θα προκύψουν ερωτήσεις για να εμβαθύνουμε σε αυτά τα ζητήματα. Ζητώ από την Επιτροπή να εστιάσει την προσοχή της σε ερωτήσεις που συνδέονται άμεσα με αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και ακούμε την κυρία Ιβάνοβα για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και επιτρέψατε μου να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετικά προσεκτική ανάλυση που κάνετε. Μας δίνει μια καλή βάση προβληματισμών, γύρει βεβαίως και πολλά προβλήματα. Ε, ε, Θεωρείται εν γέννη ότι οι φυστάμενοι μηχανισμοί του προπολογισμού για το FSM και το ESM είναι επαρκείς και διασφαλίζουν αρκετή διαφάνεια ε, για τα δύο αυτά εργαλεία, δεδομένου ότι οι συμφωνίες για το EFSM έχουν ολοκληρωθεί, αλλά το, η σύντηση για το ESM βρίσκεται υπό εξέλιξη. Ποιο είναι κατά την άποψή σα ο καλύτερο τρόπο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιφέρει κάποια προσθέμενη αξία όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο και τον ειδικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ε, άσκηση δημοκρατικού ελέγχου. Μπορείτε παρακαλώ να πάρετε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρθηκε στην ε, παρουσίαση και στην έκθεση, νομίζω ότι για το EFSM η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη υπό την έννοια ότι οι συναλλαγές του EFSM ε, ε, αναφέρονται σε αιτήσιους λογαριασμούς άρα υπάρχει δυνατότητα άσκηση άμεσου δημοκρατικού ελέγχου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ίδιο ισχύει για το συζύγιο πληρωμιο, πληρωμών και όπως αναφέρθηκε στην ε, έκθεσή μας ε, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες ε, παρατηρήσεις. Όσον αφορά δε το ESM, όπως αναφέρθηκε ήδη, το ESM στην πραγματικότητα οι συναλλαγές θα αναφέρονται, θα δηλώνονται σε μια, σε ένα, σε μια διακυβερνητική θεσμική οντότητα η οποία βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντίκτυπος στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα είναι πολύ περιορισμένος. Εκτός ε, αν κάποια, κάποιες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια κονδύλια ε, υπάρξουν, άρα θα συμπεριληφθούν σε τέτοιους λογαριασμούς η Κομισιόν και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα παρεμβαίνει έμεσα στη λειτουργία του ESM. Άρα από μια καθαρά ελεγκτική άποψη το ελεγκτικό συνέδριο με τον τρόπο αυτό θα βρίσκεται σε θέση να επαληθεύει ε, τις δαπάνες ε, και τα έξοδα και την ε, λειτουργία της Κομισιόν και των άλλων θεσμικών οργάνων όσον αφορά το ESM. Βεβαίως ε, γίνεται εκτεταμένη συζήτηση σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στη διαδικασία αυτή, καθώς ε, και για το ρόλο των ανώτατων ελεγκτικών θεσμικών οργάνων, των SAI. Νομίζω όμως ότι τελικά θα πρέπει να το δούμε. Ε, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και τα νότια ελεκτικά θεσμικά όργανα ασφαλώς ε, θα διαδραματίσουν ένα ελεγκτικό ρόλο στην αφορά στο ESM γιατί θα είναι μέλη του ελεγκτικού συμβουλίου άρα θα ελέγχουν τόσο τον εσωτερικό έλεγχο όσο και τους εξωτερικούς ελεγκτές θα παρακολουθούν το έργο τους άρα υπάρχει συμμετοχή από αυτή την έννοια επίσης οι αιτήσιοι ολοκληρωμένοι λογαριασμοί ενωπημένοι λογαριασμοί θα διαβιβάζονται ε, στους, ε, στο ελεγκτικό συνέδριο και στα εθνικά κοινοβούλια. Άρα έμεσα θα διενεργείται κάποιος έλεγχος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν τρεις άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Καταρχήν ο κύριος ε, Γιάν Μούλτερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο δημοκρατικός έλεγχος δεν μου είναι ξεκάθαρος. Όταν μιλάμε για 60 δις, τα οποία προέρχονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αποφασίζεται βάσει των συνθήκων, εγκρίνεται από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Αλλά αυτό που ακούω από την Price Waterhouse Cooper είναι ότι το Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται γιατί αλλά αυτό δεν, δεν θα ενημερώνεται μένα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο στη συναπόφαση. Και πώς θα μπορεί να αποφασίζει για την, τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα 60 δις. Απάντηση. Α, όχι, ο Πρόεδρος. Είναι δυνατόν να συγκεντρώσουμε τρεις ερωτήσεις για να απαντηθούν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε δύο επιπρόσθετες ερωτήσεις στην ε, μελέτη που κάνατε. Εξετάσατε τη νομική βάση για αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σόρεν, συγγνώμη, σε διέκοψα. Τι να κάνω, ξαναρχίσω. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η νομική βάση για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό δημοσιονομική σταθερότητα, στο EFSM, στο άρθρο 122 της συνθήκης υπάρχει μία αναφορά και θα ήθελα να ξέρω αν τη λάβατε υπόψη και αν επαρκεί η μνή αυτή ως νομική βάση για αυτό τον μηχανισμό. Άρθρο 122. Δεύτερη ερώτηση. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια πιο ρεαλιστική αξιολόγηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στα εθνικά ε, κοινοβούλια ως προς τον έλεγχο του μηχανισμού αυτού. Με ποιο τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό έλεγχο από πλευράς των εθνικών κοινοβουλίων για το ESM. Είναι δυνατό κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη σας μπορούμε να έχουμε μια συνολικότερη άποψη της κατάστασης, ε, διότι γνωρίζουμε την κατάσταση τμηματικά. Ποιες είναι οι ουσιαστικές δυνατότητες ε, που θα έχουν τα Εθνικά Κοινοβούλια για τον έλεγχο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος κυρία Ανδρέασον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία για το EFSM. Θα ελέγξει κανείς το EFSM στο τέλος της διαρκείας του. Είπατε, εν συντομία, ότι θα πρέπει να δοθούν αφορά τα εκκρεμούντα δάνεια. Όλα τα οικονομικά μέσα θα πρέπει να ελέγχονται στο τέλος των κύκλων τους. Και δεν αναφέρθηκε κάτι πάνω σε αυτό. Όσον αφορά το ESM, είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο θα έχει ένα ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο των λειτουργιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το ESM, το εξηγείτε. Και τι θα έπρεπε να ελέγχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευρύ φάσμα ερωτήσεων, λέει ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, κύριε Σονκάρ, να δώσετε απάντηση. Ο Σονκάρ. Ναι. Είναι αρκετά λεπτομερείς οι ερωτήσεις, αλλά τέλος πάντων. Ουδέν πρόβλημα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ντίρικ Βεντερίγκε, ο οποίος αναμίχθηκε και να προσθέσω τα σχόλιά μου. Για το πρώτο ερώτημα, από ό,τι κατάλαβα, αυτό θυμίζει αυτό που παρουσίασε και ο Σανκάρ στη διαφάνεια. Ρόλοι και ευθύνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το FSM ενημερώνεται μόνο για την απόφαση χορηγήσεων και δεν έχει ρόλο στην απόφαση αυτή καθ' αυτή το Κοινοβούλιο. Αυτό το σημειώσαμε. Είδαμε επίσης ότι για το MFA ότι όταν δεν επικρατούν συνθήκες ε, κατεπίγουσες μπορεί να υπάρξει συναπόφαση. Αυτά περιγράφονται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πώς λειτουργούν τα εθνικά κοινοβούλια. Και ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο ESM η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ελέγχεται μόνο από το ECAP και όχι από τους ανώτατους ηλεκτρικούς φορείς των κρατών μελών. Υπάρχει και κάποια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών για ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό μπορεί να προωθηθεί για καλύτερο, καλύτερες ελεγκτικές δυνατότητες. Τόσο αφορά το EFSM και τα εκρεμή δάνεια. Το ΙΚΑ ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα ξεκινήσουν ελέγχους για το EFSM ή ξεκίνησαν ή ξεκινάνε όπου να είναι. Θα το εξετάσουν το θέμα. Τέλος. Ποια ήταν η τελευταία ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ESM. Α, μάλιστα. Ο ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνδέεται με την αιρεσιμότητα. Ξεκινάνε με ένα μνημόνιο σε συνεννόηση με το κάτω μέλος και ελέγχουν την τήρηση των όρων κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομες ακριβείς απαντήσεις. Περνά ο χρόνος και τέθησαν ερωτήσεις που πιθανότατα μπορούν να απαντήσουν οι επόμενοι ομιλητές του πάνελ. Εγώ προτείνω να προχωρήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Άνεφ, Γενικό Γραμματέα του EFSF. Κύριε Άνεφ, καλώς ήρθατε. Ο Σεφ είναι χαρά μας που είστε εδώ και μπορείτε να πάρετε το λόγο και να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Επιτρέψτε μου καταρχάς uh, για την πρόσκληση να παραστώ σε αυτή την ακρόση και ο Ροφ Στράουχ είναι διευθυντή έρευνας και θεσμικών σχέσεων. συνάδελφο, ελπίζω και οι δύο να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Α θέσω το πλαίσιο. Όπως είπατε και αναφέρατε στην έκταση, δεν υπάρχει επίσημο δικαίωμα ή άμεση υποχρέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι του EFSF και του ESM, όμως από ευγένεια το κάνουμε αυτό εθελοντικά, ανεπίσημα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Και θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί γίνεται και όσο πιο διαφανείς γίνεται. Και ελπίζω να το σεβαστείτε αυτό. Ετοιμάσαμε μια παρουσίαση που ελπίζουμε ότι θα είδατε. Θέλω να αναφερθώ στα σημαντικότερα σημεία αυτής και να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις μετά. Σελίς 1. Βλέπετε το Σύμφωνο χρηματοσυντικής σταθερότητα που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2010. Έχουμε 60 δις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοσυντικής σταθερότητα, του FSM, η FSF με 140 δις και δούνου του 250 δις. Η εντολή μας αφορά τα 440 δις, ήταν το αρχικό πακέτο, αυξήθηκε, αυξήθηκαν οι εγγυήσεις και θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα σε σελίς 2. Το πλαίσιο βλέπετε εδώ. Ιούνιο 2010 άρχισε να λειτουργεί πλήρως το FSF και από τις 4 Αυγούστου είχαμε επαρκή υποστήριξη από τις χώρες για να δραστηριοποιηθούμε και δημιουργήθηκε το FSF σαν ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβούργου, διε, λοιπόν, μας, ε, στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου του ε, Λουξεμβούργου έχουμε ε, μετόχους, σαν μετόχους τα 17 κάτι μελη της Ευρωζώνης. Και στο Δικαιωτικό Συμβούλιο έχουμε, τους γενικού, έχουμε γενικούς ε, υφυπουργούς ε, των διαφόρων κρατών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επικεφαλής είναι ο Κλάους Ρέγκλινγκ, πρώην Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάμε στις σελίδες 3 και 4 όπου βλέπετε τι γίνεται με τους μετόχους, χώρες, κατανομή. Στη σελίδα 4 εντολές που μας ανατέθησαν, αλλά νομίζω ότι αυτά καλύφθηκαν και στην έκθεση, οπότε θα τα άφηνα εκτός αυτού και σε εστιαστούμε σε αυτά που αναφέρονται από τη σελίδα 5 και πέρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό, υποβολή αναφορών και εσωτερικό έλεγχο. Ξεκινώντας λοιπόν με τη διαδικασία του προπολογισμού, ακολουθήσαμε τη βέλτιστη πρακτική του ιδιωτικού τομέα και προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού τι γίνεται στο δημόσιο τομέα, εμπειρίες από εκεί, για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και να υποστηρίξουμε και τους ε, μετόχους μας ε, για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα χρήματα και για να υπάρχει και επαρκής ε, δημοσιονομικός έλεγχος. Παρουσιάζουμε τον προϋπολογισμό μας όπως κάθε εταιρεία ή οικονομικός φορέας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο τέλος κάθε έτους, εγκρίνεται και δίνουν ένα προσατολισμό για τον επόμενο χρόνο. Αν υπάρχουν προσαρμογές, διορθώσει για τον προπολογισμό, επιστρέφουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ζητούμε από τους αρμοδίους να εγκρίνουν ή να απορρίψουν. Μηνία γίνεται ένας έλεγχος με τους διοικητικούς φορείς και τους διάφορους αρμοδίους οι οποίοι ελέγχουν τα, τους λογαριασμούς αναλύουν τις διαφοροποίησεις και βλέπουμε κατά πόσο όλα πηγαίνουν ως έπρεπε. Ενημερώνουμε μετά καθημερινά σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν, επενδύσεις, λογιστικά, διαχείριση κινδύνου, ανάληψη υποχρεώσεων κλπ. Είναι όλες οι διαδικασίες χρηματοδότησης αυτές. Αν δούμε τι γίνεται με τον εξωτερικό έλεγχο, ακολουθούμε το IFRS, είμαστε εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο και ακολουθούμε στο μέτρο του δυνατού τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν και άλλοι διεθνείς χρηματοστηρικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμησης και Επενδύσεων και άλλοι γενικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως είναι επενδυτές και τράπεζες. Το κάνουμε αυτό διότι πρέπει να επιλέξουμε ε, σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβούργου λογιστικά πρότυπα και αυτό είναι κάτι που συμφέρει και τους επενδυτές μας. Για να συλλέξουμε τα ποσά πάμε στις αγορές κεφαλαίων και πρέπει οι επενδυτές να καταλάβουν πώς είναι οι λογαριασμοί μας και ξέρουν τα ΕΦΡΕΣ, τα πρότυπα αυτά που χρησιμοποιούνται από διάφορους χρηματοσυντικούς φορείς. Καλύπτονται λοιπόν τα περισσότερα γενικά θέματα έλεγχο λογιστικών, διαδικασίε συναλλαγών, έλεγχη, πολιτικέ διαχείριση κινδύνων, που είναι σημαντικό θέμα. Ενημερώνουμε και υποβάλλουμε αναφορέ όχι μόνο μία φορά το χρόνο, που είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με τον νόμο του Λουξεμβουργού, και εγκρίνεται η αναφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκεί συμμετέχουν 17 κράτη-μέλη, αλλά εθελοντικά υποβάλλουμε αναφορέ και στέλνουμε αιτήσει λογαριασμού που ελέγχονται από το PwC. Το διαλέξαμε αυτό εδώ, αυτόν τον τρόπο εδώ και δύο χρόνια. Υποβολή αναφορών σε εξωτερικούς φορείς, ποιότητα στατιστικών στοιχείων, κάτι που αναφέρεται στην έκθεση. Να σας δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Ξεπερνούμε αυτό που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο του Λουξεμβουργού ε, υποβάλλουμε αναφορές στην Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου και Στατιστική Υπηρεσία του Λουξεμβούργου και στη Eurostat ε, κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο και κάθε χρόνο, όχι υποχρεωτικά, θελοντικά. Αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Και για να γίνει αυτό και διάφορες στατιστικές ε, ε υπηρεσίες να μπορούν να ενημερώνουν και τις αρμόδιες φορείς των κρατών μελών. Στη σελίδα 9 και 10 Καλύπτουμε τον εσωτερικό έλεγχο, θα επιστρέψω σε λεπτομέρειες. Έχουμε όμως εσωτερικό έλεγχο. Δεν είναι υποχρεωτικό νομικά, το κάνουμε, διότι πιστεύουμε ότι είναι καλό για τον οργανισμό μας. Χρειάζεται εσωτερικός έλεγχος, ανεξάρτητος, που μπορεί να επικρίνει επικοδομητικά τυχόν λάθη, να μπορεί να επιφέρει βελτιώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ως οργανισμό και μπορούμε να βοηθήσουμε και τους ανώτερους αρμοδίους φορείς μέσω του κεντρικού ελέγχου να πετύχουμε εξάρτητο έλεγχο. Και υπάρχει και επαφή με τους ελεγκτικούς φορείς και το Διοικητικό Συμβούλιο για να δικαιολογούνται αποφάσεις που ελήφθησαν ή για να εντοπίζονται σημεία μια Σελίδα 11. Αναφερόμαστε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας βασικό θέμα που θέλετε να συζητήσουμε, όπως αναφέρθηκε σωστά από τους προλαλήσαντες, το ESM είναι διακυβερνητικό φορέας που διέπεται από διεθνέ δίκαιο. Δεν είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσης, ούτε ιδιωτική εταιρεία όπως το EFSF. Δανειοδοσία πάει μέχρι 500 δις, 700 δις κεφάλαιο 80 δι από αυτά θα καταβάλουν και 680 θα, είναι, θα συλλέγονται η διακυβέρνηση, η είναι διαφορετική, διοικητικό συμβούλιο και από πάνω είναι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, 17 χώρες για την ώρα. Και έχουμε το Διευθυντικό Συμβούλιο που είναι το ίδιο όπως το EFSF, συνδυάζουν διευθυντέ και θα συμμετέχουν και τα μέλη, κράτη-μέλη του Eurogroup. Υφυπουργοί Οικονομικών, ε, γενικοί διευθυντέ και διάφοροι αρμόδιοι των κρατών μελών. Μετά έχουμε το Διευθυντή όπου διαχειρίζεται εσωτερικά θέματα του ESM. Έχουμε το ελεκτικό συνέδριο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και με εθνικούς ελεγκτικούς φορείς για να γίνεται σωστός έλεγχος για το ESM και για τη διεξαγωγή συζητήσεων. Αποτέλεσμα αυτού Διορίζονται πέντε μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο που θα είναι στο ε, ελεγκτικό συνέδριό μας. Ένας θα διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, δύο από τα εθνικά ελεκτικά όργανα και δύο ανεξάρτητοι πυρογνώμονε. Αυτό συνάδει με τη βέλτιστη πρακτική άλλων φορέων. Εξετάσαμε τι γίνεται με το Δουνουτίου και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμηση και Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εξετάσαμε τι γίνεται με άλλους παρόμοιους φορείς και να δημιουργήσουμε μια δομή συγκρίσιμη. Σελίδα 13. Εξηγούμε πώς το FSF και το ESM θα τρέχουν παράλληλα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό τώρα, δεν είναι σημερινό θέμα. Θα εστιαστώ στη σελίδα 14 όπου προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τα άρθρα συνθήκης ESM που αναφέρονται στον προπολογισμό και τους ετήσιους λογαριασμούς, εσωτερικό, εξωτερικό έλεγχο, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος τώρα γίνεται βάσει βέλτιστης πρακτικής. Προσπαθούμε να πετύχουμε διαφάνεια στο βαθμό του δυνατού δημοσιεύουμε τις εκθέσεις στην ιστοσελίδα μας. Αυτό αναφέρθηκε και στην έκθεση. Εδώ θέλουμε να επιτεθεί μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Σελίς 15. Εκεί αναφέρεται το ελεκτικό μας συνέδριο, φορές τον ο ελεγκτικός, τι δικαιοδοσία έχουν και αυτά στις λεπτομερείς διατάξεις του ΕΣΕΜ αναφέρονται. Σελίδα 16 βλέπουμε τις συζητήσεις που διεξάγονται τώρα με τα κράτη-μέλη, τα βασικά σημεία. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω για την ώρα. Βρισκόμαστε το μέσο συζητήσεων με τα 17 κράτη-μέλη. Έχουν προταθεί διάφορα κείμενα για το πώς θα η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πώς θα διορίζονται τα μέλη, ποια είναι η αρμοδιότητα του ελεκτικού φορέα κλπ. Πώ θα λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και αν θα υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων με το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι λεπτομερεί διατάξει θετηθούν. Ο εσωτερικό κανονισμό θα θετηθεί τον Ιούλιο του 2012, όταν θα έχει συσταθεί επίσημα το ESM. Για την ώρα διεξάγονται συζητήσει, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε εσωτερικό κανονισμό διατάξει οι οποίε θα τύχουν υποστήριξη και θα αντικατοπτρίζουν τι ευθύνε όλων των συμμετοχόντων εδώ θα σταματήσω. Στη σελίδα 17 το EFSF ιδρύθηκε σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις των κρατών, υιοθετήσε το Άφερες που αναφέρεται στον έλεγχο, λογιστικά, διαχείριση κινδύνου Εθελοντικά έχουμε καθορίσει βέλτιστες πρακτικές πέραν των υποχρεωτικών όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Εθελοντικά έχουμε καθορίσει αστασιακά στοιχεία, εξωτερικό έλεγχο, υποβολή αναφορών, σημαντικά όλα αυτά για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών και για το ESM θέλουμε να δημιουργήσουμε υποδειγματικό φορέα μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και ε, ε, του εσωτερικού κανονισμού, άμα όλα αυτά ετοιμαστούν, θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες και ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα υποδειγματικό φορέα. Ευχαριστώ κύριε Άνεφ. Για, αυτή την, για αυτά τα εισαγωγικά σας λόγια υπάρχουν καθόλου ερωτήσεις από το πάνελ. Κυρία Ιβάνοβα, συγγνώμη, νομίζω ότι βιάστηκα. Θα, το, θα συζητήσουμε τις δύο παρουσιάσεις από κοινού θα το συζητήσουμε μαζί με, ε, με την παρουσίαση του κυρίου Μπούτη. Ευχαριστώ πολύ. Και καλώς ήρθατε κύριε Μπούτη για να μας παρουσιάσετε το άλλο τμήμα της προβληματικής αυτής. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Δεν είμαι τακτικός ε, επισκέπτης σε αυτή την επιτροπή, συνήθως πάω στην ΕΚΟΝ αλλά είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Και επιτρέψατε μου επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ιβάνοβα για την έκθεσή της και επίσης ε, το, την PwC, ε, την Price ε, Waterhouse, Waterhouse Cooper, η οποία για τη μελέτη της είναι νομίζω συμπληρωματική η αξία της γιατί θέτει πολύ σημαντικά ζητήματα για το EFSF και το ESM. Όπως ε, αναφέρθηκε ήδη το EFSM δημιουργήθηκε βάσει του κανονισμού 407 κάθετος 2010 που δίνει στην Επιτροπή το δικαίωμα να, κεφανί... να δανείζεται χρήματα από τις κεφαλαγορές και να δανείζει τα χρήματα αυτά σε μια χώρα μέλη μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολία. Και επειδή τα δάνεια υπό την του FSM υποστηρίζονται από τον προπολισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγχει τι ενέργειε τη Επιτροπή όσον αφορά το EFSM και επίση μπορεί να διενεργεί έλεγχο για, τις, για τη λειτουργία τη Επιτροπή στο πλαίσιο του προπολογισμού και τη διαδικασία τη απαλλαγή. Και αναφέρθηκε προηγουμένω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει άμεση δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Και αυτό αφορά την νομική βάση, δηλαδή το άρθρο 122. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δικαιώματα, πλήρη δικαιώματα ελέγχου για το πρόγραμμα αυτό, καθώς για όλες τις ε, δανειοληπτικές και δανειοδοτικές δραστηριότητες της Επιτροπής και για το EFSM. Άρα το συμπέρασμα είναι το IFSM υπόκειται σε έναν επαρκή δημόσιο έλεγχο και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, το IFSM είναι ένα εργαλείο της Ένωσης, γι' αυτό υπόκειται στο γενικό πλαίσιο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βάσει το οποίο επιτροπή είναι πάντοτε υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κατά τη με το BOP και το MFA, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει πλήρη ελεγκτική πρόσβαση όσον αφορά το EFSM. Επίσης, όσον αφορά το ΙΕΦΣΜ, ο ειδικό του ρόλος τονίζεται στο άρθρο 3.5 του κανονισμού, όπου λέει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διαβιβάζει το μνημόνιο στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε χώρα που παίρνει δάνειο υπό του BOP ή του EFSM ε, γίνεται κάθε τρίμηνο μια αξιολόγηση όσον αφορά την εκπλήρωση των όρων πριν εκταμιευθεί η επόμενη δόση. Και αυτές οι εκθέσεις δημοσιεύονται και διαβάζονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης γίνονται τακτές εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά τη δανειοληπτική και δινεδυτική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για τις εγγύησεις που καλύπτονται από το προπολογισμό. Ως εκ τούτου η Επιτροπή πάντοτε παρέχει επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τις δανειοληπτικές και δινεδυτικές δραστηριότητες. Επίσης αναφέρονται και υποβάλλονται σε έλεγχο στους ετήσιους λογαριασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο μέσω της έγκρισης του προπολογισμού και της διαδικασίας απαλλαγής. Ε, συνολικά η Επιτροπή θεωρεί ότι το πλαίσιο του EFSM και η ανάθεση ρόλων και ευθυνών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων είναι απολύτως ανταδειγμένη. Υπάρχουν βεβαίω κάποια ουσιαστικά μέτρα ώστε να διαφυλάξουν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ομόλογα τα οποία εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δάνεια αυτά γίνονται σε ευρώ Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ανοιχτά επιτόκια ή δεν υπάρχουν προβλήματα στον αφορά τι συναλλαγματικές ισοτιμίες και αυτό γίνεται για να προστατεύει το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η αποπληρωμή εκ μέρους των χωρών ε, φροντίζει για τα ομόλογα, την κάλυψη των ομολόγων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ε, περίπτωση χρεοκοπίας, η διαχείριση των, της ρευστότητας εκ μέρους της Επιτροπής και το δικαίωμα της Επιτροπής να αντλήσει χρήματα από τις εισφορές των χωρών εξασφαλίζει μια έγκαιρη αποπληρωμή όλων των υποχρεωτικών δαπανών ε, συμπεριλαμβανόμενης και της εξυπηρέτησης του χρέους για τα ομόλογα τα οποία εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει μια πρόταση για ένα διορθωτικό προπολογισμό ούτως ώστε να λογοδοτήσει για αυτά τα ποσά ε, στον, στην αντίστοιχη γραμμή του προπολογισμού που αφορά το EFSM. Ε, το IFSF και το ESM είναι δύο μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής συνδρομής οι οποίοι δημιουργήθηκαν ως ανεξάρτητες οντότητες μέσω μιας συμφωνίας ή μιας διεθνούς συνθήκης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και ε, βρίσκονται εκτός του πλαισίου της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δανειοδοτικές δραστηριότητε υποστηρίζονται πλήρως από τις χώρες μέλη και δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει έναν κρίσιμο ρόλο, ο οποίος εδράζεται στη συνθήκη για το ESM είναι υπεύθυνη η Επιτροπή για να διαπραγματεύεται της, ε, την αιρεσιμότητα η οποία συνδέεται με την παροχή χρηματοοικονομικής συνδρομής και την παρακολούθηση της, ε, της εκπλήρωσης αυτών των όρων. Κάθε χώρα η οποία δέχεται χρηματοοικονομική συνδρομή υπό την αιγίδα του EFSF ή του ESM θα υπόκειται σε τακτές αξιολογήσεις όσον αφορά την εκπλήρωση των όρων που έχουν τεθεί. Στην περίπτωση δανείων, τέτοιου είδους αξιολογήσεις γίνονται κάθε τρίμηνο και πρέπει να ολοκληρωθούν πριν εκταμιευτεί η επόμενη δόση. Ε, όλες αυτές οι, εκδόσεις, οι εκθέσεις συγγνώμη, δημοσιεύονται ε, και τα μνημόνια τα οποία υπογράφουν στις χώρες αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως συνέβη στην περίπτωση της ε, οικονομικής συνδρομής υπό την αιγίδα του EFSF. Ε, πέρα από αυτό θα ήθελα να τονίσω ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο κανονισμό ε, το, υπό το άρθρο 136 το οποίο αποσκοπεί να εξασφαλίσει μια συνέπεια μεταξύ των διαδικασιών που ε, εγκαθιδρύονται υπό το πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο για το AFSF και για τη συνθήκη του ESM και το πλαίσιο πολυμερούς παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, αυτό είναι αντικείμενο συνεξόμενης διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμπίπτει στην απόφαση. Άρα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει ένα πλήρη ρόλο όσον αφορά την έγκριση αυτή τη συμφωνία. Όσον αφορά τη λογοδοσία για το EFSF και το ESM, έχει γίνει σημαντική εργασία για να εξασφαλίσει όχι μόνο τη διαφάνεια αλλά και τη λογοδοσία για το EFSF και το ESM, παρόλο που υφίστανται εκτός του πλαισίου της συνθήκης. Καταρχήν, το EFSF ε, προβλέπει κάποιες διευθετήσεις όσον αφορά την εξασφάλιση του δημόσιου εξωτερικού ελέγχου και σαν ε, μια εταιρεία η οποία έχει την έδρα στο Λουξεμβούργο υπόκειται στις νομικές διατάξεις του Λουξεμβούργου σαν αφορά τη διενέργεια ελέγχων ε, και προβλέπεται ότι θα πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι λογιστές ε, οι οποίοι θα ψηφίσουν από τους μετόχους για μια μέγιστη διάρκεια 6 ετών. Αυτοί οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητα εξωτερικοί, εξωτερικοί ελεγκτές, αυτή τη στιγμή είναι το PwC και επιπρόσθετα το EFSF προβλέπει μια εσωτερική διαδικασία ελέγχου την οποία παρουσίασε ο συνάδελφος προηγουμένως. Επειδή το ESM είναι ένας μόνιμος μηχανισμός, ε, έχει προπάρξει συνεργασία με τις ανώτερες ελεγκτικές αρχές, ούτως ώστε να αναπτυχθεί μια διαδικασία ελέγχου η οποία να προβλέπει για τις βέλτιστες πρακτικές και να τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές. Ε, και η διατάξη σχέση με τον έλεγχο ε, για, ε, στο πλαίσιο της συνθήκης του ESM ε, συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών ελέγχου που προβλέπονται για αντίστοιχους ε, παρόχους ε, οικονομικών, δημοσίους παρόχους οικονομικών υπηρεσιών. Το ESM θα περιλαμβάνει τρία επίπεδα ελέγχου, έναν ιστορικό έλεγχο, έναν εξωτερικό ανεξάρτητο έλεγχο και έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό συμβούλιο. Το ελεγκτικό συμβούλιο θα έχει την δυνατότητα να διενεργεί ανεξάρτητους ελέγχους σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, και η αιτήσια του έκθεση θα είναι προσιτή από τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις ανώτες εποπτικές αρχές των μελών του ESM και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διαφάνεια και οι λεπτομερείς διατάξεις για το ESM όσον αφορά τον έλεγχο έχουν ε, ήδη ε, προπαρασκευαστεί περιλαμβάνοντας ε, ε, την γνώμη την οποία έχουν εκδώσει ανώτατες εποπτικές αρχές και έχουν εγκριθεί πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Στις ε, συναντήσεις ε, της Άνοιξης με το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανέκυψαν κάποια προβλήματα και μας επέκριναν ότι ε, δεν ε, βάζουμε αρκετά χρήματα στο EFSF, στο ESM, στο FSM κλπ. Ε, αυτό το οποίο συζητούμε εδώ δείχνει ωστόσο ότι έχουν δεσμευτεί μεγάλα ποσά για να προστατευτεί η σταθερότητα της Ευρωζώνης και του ευρώ. Αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι προσπαθήσαμε και πραγματικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε ε, ούτως ώστε πέρα από την κινητοποίηση αυτών των χρηματικών πηγών προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 60 δις για το ESM υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη το αναγκαίο περιθώριο ε, το υφιστάμενο μάλλον περιθώριο ελιγμών ούτως ώστε η δύναμη πυρός να κεντοποιηθεί μόνο σε καταστροφικές ε, περιστάσεις κατακλυσμιές ε, φύσης η χαρακτήρα. Άρα λοιπόν έχει διασφαλιστεί εδώ η πλήρης προστασία. Και ένα δεύτερο σημείο αφορά το εξής. Όλο αυτό το οικοδόμημα δεν ήταν ε, μια, ένα εύκολο εγχείρημα για τα θεσμικά οργάνα της Ένωσης. Το Μάιο του 2010 όταν ε, δημιουργήθηκε το EFSF και το FSM προτείναμε κοινοτικά όργανα. Αλλά το Συμβούλιο εκείνη την εποχή ε, δεν συμφώνησε με αυτή την άποψη και συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί το FSM ε, κάτω από το κοινοτικό πλαίσιο και το SM εκτός. Ε, γιατί πρόκειται για μια διακυβερνητική συνθήκη. Άρα ήταν κάπως ευαίσθητο το σημείο αυτό όσον αφορά την Επιτροπή και το ρόλο που καλείται να παίξει. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια τη συζήτηση είναι να ευθυγραμμίσουμε ή δυνατόν τις απαιτήσει, τι διαδικασίε καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των εργαλείων συμβάλλοντα σε αυτή τη συζήτηση με τι διαδικασίε και την προσέγγιση η οποία ε, κυριαρχεί και εμπίπτει στην ε, κοινοτική μέθοδο και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Και ε, όπως σας είπα προτάθηκε κανονισμός που προβλέπει την απόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μιας συνέπειας, μιας συνοχής λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι το ESM το οποίο τον Ιούλιο του 2012 ε, θα λάβει τα ε, σκύπτρα θα παραμείνει υπό την αιγίδα της ε, διακυβέρνησης. Πρόκειται λοιπόν για μια συνεχιζόμενη και συνεχή προσπάθεια και ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο από θεσμική άποψη και διατυπώσαμε κάποιους ε, κανόνες για αιρεσιμότητα που να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την ε, πολυτερημερή παρακολούθηση και το Sixth Pack και στην πρόταση του νέου κανονισμού που βρίσκεται τώρα υπό συζήτηση. Και επίσης ε, προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να το κάναμε διατυπώσαμε κάποιες ε, αρχές για την παρακολούθηση ε, στη συνέχεια ούτως ώστε να συμπεριλάβουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις χώρες μέλη όχι μόνο κατά την ίδια την ε, περίοδο εφαρμογή του προγράμματος όπου υπάρχει αυστηρή τήρηση των όρων, αλλά και στην περίοδο που ακολουθεί. Αυτά λοιπόν ε, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσπάθειάς μας. Και δεν μπορώ παρά να απευθύνω μία έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το Συμβούλιο, ούτως ώστε να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατό την πρόταση υπό το άρθρο 136 που θα ενισχύσει ακριβώς το ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων όσον αφορά τη δύναμη πυρός και των χωρών στόχος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάρκο Μπούτη. Ε, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΚΦΙΝ, σας καλωσορίζουμε και πάλι. Ε, μία ερώτηση διευκρινιστική. Αντελήφθη ορθά αυτό που είπατε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον ESM ότι προς το παρόν είναι πολύ πιο αδύναμο σε σχέση με τον προηγούμενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του EFSM. Κατάλαβα καλά ότι όπως έχουν τώρα τα πράγματα ο ρόλος της Επιτροπής στο ESM είναι πολύ ασθενέστερο σε σχέση με τον προηγούμενο ρόλο που είχε στο EFSM. Απάντηση. Ως προς την εφαρμογή ε, της αιρεσιμότητας και την ε, διαπραγμάτευση του Μνημονίου Συνεννόησης ε, είναι ίδιος και απαράλλαχτος ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν μιλάμε δηλαδή για την εποπτεία των εθνικών προγραμμάτων. Για την Το EFSM, το EFSF και το ESM έχουν, υπακούν μάλλον στον ίδιο κανόνα. Στο EFSM Βεβαίως είμαστε απολύτως υπεύθυνοι για την δανειοδοτική και δανειοληπτική δραστηριότητα βάσει του προϋπολογισμού. Αυτό δεν ισχύει ούτε για το EFSF ούτε για το ESM. Η επόμενη ερώτηση του κυρίου Τόιρερ Ποιος είναι υπεύθυνος λοιπόν η... το διακυβερνητικό διοικητικό συμβούλιο, ποιος είναι αρμόδιος στο ESM για τη δανειοδότηση. Εφόσον με ρωτάτε κάτι για το ESM, είναι προφανές ότι καλύτερα θα ήταν να απαντήσουν οι συνάδελφοι. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η Υπουργή Οικονομικών ουσιαστικά των κρατών το λειτουργικό του βραχίωνα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως προαναφέραμε, που έχει ε, εξουσιοδότηση, έχει λάβει εντολή για αυτά τα ζητήματα. Για τη δανειοδοτική και δανειοληπτική δραστηριότητα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλιστα, λέει ο κύριος Στόιρερ. Θέλετε κι εσείς να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Μπούτη. Αληθεύουν, πρόκειται για μια διακρατική οργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα του Διοικητικού Συμβουλίου. Εξουσιοδοτείται ο εκτελεστικός διευθυντής επίσης να εξ ονόματος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Ιβάνοβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους ε, προλαλήσαντες ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του EFSF. Αδειμονώ για την παρέμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά προ τον κύριο Άνευ θέλω να ρωτήσω το εξή. Η συνύπαρξη αυτών των δύο μηχανισμών, EFSF και ESM, ε, τι συνεπάγεται, δηλαδή ποιο θα υποπτεύει τον συντονισμό ανάμεσα στα δύο, γιατί είναι όχημα ε, ε, ειδικού στόχου το EFSM και θα συνεπάρχει για ένα χρόνο με το ESM. Πώ θα γίνει το συντονισμό, Δεύτερη ερώτηση που έχουμε ξανασυζητήσει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αν προκύψει bailout, διάσωση κάποιου κράτου, επί ποιε βάσει θα ληφθεί η απόφαση για να γίνει επιλογή ανάμεσα στο EFSF και το ESM. Υπάρχουν σαφή προκαθορισμένα κριτήρια σχετικά με την επιλογή ανάμεσα στα δύο όργανα κατά την περίοδο συνύπαρξή του και μια άλλη ερώτηση. Τι πιστεύετε σε σχέση με τη χορήγηση τραπεζικής άδειας στο ESM. Υπάρχουν, ε, υπάρχει, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις αυτή η ερώτηση προς ε, τον εκπρόσωπο του EFSF και προ τον κύριο Μπούτη. Ε, θέλω να ρωτήσω το εξή. Αναφερθήκατε στην παρουσίασή σα επανειλημμένα στο εξή, ότι υπό συγκεκριμένε περιστάσει ε, δεν υπάρχουν σοβαρέ δυνατότητε πτώχευση, αθέτηση υποχρεώσεων σε επίπεδο κράτου. Είμαστε καλά προστατευμένοι, μα είπατε. Εγώ έχω ενδιασμού. Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας δανειοδότης με υψηλή βαθμολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο υποβόσκον ε, ε, κίνδυνος συναλλαγών είναι υπαρκτός. Δηλαδή, οι ε, οφειλέτες ε, έχουν χαρακτηριστεί από τις αγορές ε, ως οφειλέτες υψηλού κινδύνου. Παρότι έχουμε λοιπόν δανειστές υψηλότατης ποιότητας, αν οι οφειλέτες δεν είναι εξίσου υψηλής ποιότητας, ποια κατάσταση θα δημιουργηθεί Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μιλάμε για το EFSF είτε για το ισοζύγιο πληρωμών, δεν έχουμε εγκυοδοτικό ταμείο όπως ε, στα πλαίσια του μηχανισμού MFA, μακροοικονομικής βοήθειας. Πώς λοιπόν θα προστατευτεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι ελοχεύει σοβαρά κίνδυνος σε αυτές τις ε, δραστηριότητες. would you like to start? Ε, κύριε Άνοφ, θέλετε να αρχίσετε εσείς γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Μάλιστα, ευχαριστώ. Θα απαντήσω ε, στην πρώτη ερώτηση και τις επόμενες θα τις δώσω στον συνάδελφό μου. Για το EFSF και το ESM, πώς θα λειτουργήσει ο συντονισμός αυτό τον πρώτο χρόνο που θα συνεπάρχουν. Θα έχουν την ίδια διακυβέρνηση, δηλαδή το ίδιο διοικητικό συμβούλιο θα διαχειρίζεται και το EFSF και το ESM και κατά πλειοψηφία αυτό ισχύει και για το προσωπικό που θα στελεχώνει αυτούς τους οργανισμούς. Ε, αυτό είχαμε προβλέψει. Ίδιο προσωπικό, ίδιο διοικητικό ε, συμβούλιο για τους ε, δύο οργανισμούς. Η έδρα τους θα είναι στο ίδιο κτίριο, στο Λουξεμβούργο. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι συνιστούν δύο διαφορετικές νομικές οντότητες, αλλά η διαχείριση εναπόκειται στους ίδιους φορείς. Για τις επόμενες ερωτήσεις θα ακούσουμε τον συνάδελφο. Μάλιστα. Για τη μεταβατική περίοδο θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση. Στην διαφάνεια υπερθμών 13 της παρουσίασης που έχετε λάβει δίνεται η απάντηση. Η εξαγγελία του Eurogroup πριν από τρει εβδομάδες έχει καταλητική σημασία από αυτή την άποψη. Αναφέρεται ότι οι φυστάμενε αναλήψεις υποχρεώσεων μέχρι τον Ιούλιο του 2012 θα εξυπηρετηθούν από το EFSF οι νέε από το ESM. Αν δεν συμβεί κάτι άλλο, τα τρέχοντα προγράμματα για την Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα θα συνεχίσουν να τρέχουν και να καλύπτονται από το EFSF. Αν προκύψει κάτι καινούριο, τότε ε, θα εμπλακεί το ESM και θα αναλάβει. Σχετικά με τη χορήγηση τραπεζικής αδείας ε, δεν έχει γίνει καμία τέτοια προσπάθεια ούτε για το EFSF ούτε για το ESM. Thank you very much. Mr. please. Ο κύριος Μπούτη τώρα. Yeah, thank you Σας ευχαριστώ πολύ εύστοχα τα ερωτήματα. Ε, θα ήθελα να πω ότι μόλις ε, βγήκαμε από μια περίπλοκη άσκηση αναδιάρθρωσης ε, στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν η, με, η μεγαλύτερη σε κλίμακα σε όλη την ιστορία και καταφέραμε παρόλα αυτά προστατεύσουμε όχι μόνο τον προϋπολογισμό της Ένωσης αλλά και τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τους προϋπολογισμούς των δημοσίων φορέων των κρατών της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι αυτό είναι τρανή απόδειξη ακόμη ε, και στα πλαίσια τέτοια ε, μεγάλη κλίμακα αναδιάρθρωση καταφέραμε να προστατεύσουμε τα δημόσια συμφέροντα. Δεύτερη παρατήρηση. Αναφέρθηκε με σαφήνεια και υπάρχει πλήρης δέσμευση από πλευράς ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων ότι στην περίπτωση της Ελλάδας πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν υπάρχει η πρόθεση να επαναληφθεί. Η εμπειρία αυτή ε, ελήφθη η απόφαση να υπερβούμε το δόγμα, το υπονομαζόμενο Ντοβίλ, δόγμα της Ντοβίλ δηλαδή, που έχει ενταχθεί και στη συνθήκη για τη σύσταση του ESM. Πέραν αυτού, Έχουμε δικλείδες ασφαλείας άμεσης εφαρμογής για την προστασία του προϋπολογισμού. Να σας πω πώς λειτουργεί ο μηχανισμός. Αν η εξυπηρέτηση του χρέους δεν λαμβάνεται την ημέρα ταφ 14 σε σχέση με τη μεταφορά πιστώσεων ε, του ESM ή τι μείον 7 ημέρες ε, στα πλαίσια του ισοζυγίου πληρωμών θα χρησιμοποιήσει το δικό της ταμείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν χρειαστεί θα αντλήσει εκτάκτος πόρους από τους δικούς τους πόρους προς όφελος των κρατών μελών βάσει του ισοζυγιου πληρωμων θα χρησιμοποιησει το δικο της ταμειο η ευρωπαικη επιτροπη η αν χρειαστει θα αντλησει εκτακτο πορους απο τους δικους τους πορους προς οφελος των κρατων μελων βασει του αρθρου 12.3 του κανονισμού 1150 του 2000. Εφόσον για τις πληρωμές, τα κράτη-μελή χρειάζονται τρεις ημέρες, ώστε να συμμορφωθούν με την αίτηση, το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αυτές οι 14 μέρες για το EFSF και οι 7 για το BOP θεωρείται ότι επαρκούν. Στη συνέχεια, πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού προβλέπεται ώστε ε, στη γραμμή ε, προσυπόμνηση PM του προϋπολογισμού της Ένωσης ε, για το BOP και για το EFSM να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αυτά τα κονδύλια. Υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στο EFSM και το ισοζύγιο πληρωμών, το BOP, η οποία συνδέεται με το εξή. Εφόσον για το EFSM μιλάμε για ε, δάνεια εκτός Ένωσης, η μόχλευση για την αποπληρωμή είναι προφανώς ε, χαμηλότερη σε σχέση με δάνεια που χορηγούνται ε, σε κράτη-μέλη της Ένωσης είτε εντός είτε εκτός της Ευρωζώνης. Ιδού η προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης το 9% του συνολικού ποσού είναι ε, στην, ε, ε στη γραμμή που ε, χρησιμοποιείται για τα εξωτερικά δάνεια. Το ίδιο ισχύει και για το BOP και για το IFSM. E είναι περιορισμένος ο αριθμός των ε, συμβαλωμένων μερών, ε, αυτή τη στιγμή είναι πέντε το αριθμό που εκπροσωπεί που αντιστοιχούν σε εγγύηση σε δισεκατομμυρίων ε, δεν χρειάζονται καν όλες αυτές οι εγγύησεις στην περίπτωση του EFSM. Στον ΠΟΠ τώρα, όπου αντιγράψαμε ουσιαστικά το πρότυπο του EFSM, έχουμε αυτήν την δικλίδα που σας είπα 14 ή 7 μέρες πριν τις πληρωμές έχουμε ένα περιθώριο ελιγμών και ζητάμε από τα κράτη-μέλη αν συντρέξει λόγος να ε, προτείνουν μια πιο ε, ενδεδειγμένη λύση. Αλλά πάντως τονίζω αυτό που σας είπα και στην αρχή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση να επαναληφθεί η ίδια εμπειρία όπως στην περίπτωση της ε, αναδιάρθρωσης του χρέους στην Ελλάδα και η άμεση εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση αιρεσιμότητα σε σχέση με τα άλλα εθνικά προγράμματα θα διασφαλίσει το ότι δεν θα επαναληφθεί αυτή η εμπειρία στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε. Και τώρα έχω πολλούς συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Προτείνω δύο γύρους ερωτήσεων. Και Γκολτ, Σέντεργκαρτ και Μούλτερ, πρώτος γύρος. Αντρεάσαν, Γκάιερ και Οντί στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, αλλά της Οικονομικής Επιτροπής. Uh, Έχω σύντομη ερώτηση. Πρώτη είναι για μια διευκρίνηση. Δεύτερη προς τον κύριο Μπούτι. Άκουσα με τα μεγάλης προσοχής. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα του κοινοτικού προπολογισμού. Από την άλλη, συγκρίνοντας τα ποσά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση Ιρλανδίας και Πορτογαλίας και συγκρίνω το μέγεθος των χρηματοδοτήσεων, το IFSM e 60 δισεκατομμύρια. Η FSF 440 και στη βρημένη εκδοχή 780. Πορτογαλία 26 δις EFSM, ESM και 26 EFSF και 26 του Δουνουτού. Συγκρίνεται με την Ιρλανδία, είναι παρεμφερή. 22,5 δις EFSM χρησιμοποιήθηκαν. Άρα από τα 60 δις 48,5 χρησιμοποιήθηκαν για Ιρλανδία και Πορτογαλία. Ενώ το EFSF χρησιμοποίησε πολύ λιγότερα. Διερωτώ τι γίνεται, συγκρίνοντας τώρα τα ποσά που εκταμιεύθηκαν από το FSF και βλέποντας το μερίδιο, το ποσοστό του, των χρημάτων που διακινδυνεύει, που δόθηκε από το EFSM, γιατί συγκρίνονται έτσι τα ποσά. Γιατί τα FSM, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από το EFSF. The Πώς εξηγείται αυτό και δεύτερον, ποια δράση ανελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αλλάξει το ποσοστό ούτως ώστε να είναι θετικότερο το αποτέλεσμα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Όσον στα έγγραφα που έχουμε παραλάβει από το EFSF. Όπως γράφεται λοιπόν και όπως αναφέρθηκε, βλέπουμε ότι τον Ιούλιο του 2013 θα σταματήσουν τα προγραμμάτα. Εξού και η ερώτησή μου. Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία πότε αναμένεται να καταργηθεί το EFSF, να πεθάνει, να πάψει να υφίσταται, να διαλυθεί. Δεύτερον, η έδρα στο Λουξεμβούργο είναι κάτι τεχνικής φύσεως. Υπάρχει τεχνική εξήγηση. Γιατί επελέγει το Λουξεμβούργο. Ε, Είχατε υπόψη συγκεκριμένους ελεγκτικούς κανόνες που σας έκαναν να προτιμήσετε το Λουξεμβούργο εν συγκρίση με άλλες τοποθεσίες. Κι άλλη μια ερώτηση. Σωστά κατάλαβα ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας το EFSF, τα λογιστικά, οι λογαριασμοί του EFSF ελέγχθηκαν από την, ε, ε, ε, τη, House Water Cooper. Τη Waterhouse Cooper, μάλλον. Ο Ιαν Μούλτερ στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξακολουθώ να είμαι μπερδεμένο. Το Μάιο του 2010, με υπό την πίεση τη χρονική, μέσα άνοιχτα και ανοίγοντα τα χρηματιστήρια στο Τόκιο, πάει σε απόφαση και δεσμεύει 60 δι του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού από το EFSM. Εντάξει, υπήρχαν πίεσει. Αλλά η εξήγηση του κυρίου Μπούτι δεν είναι σαφή. Σύμφωνα με τη συνθήκη, το Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζουν για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Τώρα επενδύουμε τα χρήματα τα 60 δις, χρησιμοποιούμε τα χρήματα και τώρα μου λένε ότι από τα 60 δις που είναι το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί κάποια νομική βάσεως έχει μόνο το δικαίωμα ενημέρωσης. Πώς γίνεται αυτό. Ερμηνεύω εσφαλμένα τη συνθήκη, κάτι συμβαίνει με το μυαλό μου, τον τρόπο σκέψης μου. Θα ήμουν ευγνώμων αν ελάμβανα μια σαφή απάντηση από τον κύριο Μπούτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος μπορεί να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα των απαντήσεων. Τα περισσότερα ερωτήματα απευθύνθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι και έτσι τα πράγματα. Ποιος μπορεί να ξεκινήσει. Ορίστε. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο για τις ερωτήσεις. Αυτές που απευθύνθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρχάς. Γίνεται γενικός επιμερισμός μεταξύ χρημάτων ευρωπαϊκών και δούνου του στα προγράμματα. Στα αρχικά προγράμματα, δύο τρίτα, ένα τρίτο ήταν το μοίρασμα. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελλάδας άλλαξε κάπως για διάφορους λόγους. Αν θέλετε μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιραστήκανε μεταξύ FSM και FSF. Γιατί το μερτικό του FSM είναι μεγαλύτερο στα αρχικά προγράμματα από ότι το EFSF. Για δύο λόγους βασικά. Πρώτον, το EFSF ήταν εντελώς καινούριο θεσμός. Έπρεπε να συσταθεί εν πρώτης. Οπότε η δανειοληπτική και η δανειοδοτική διεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε, το κάναμε για τα MFA, από την αρχή της κρίσης με το BOP. Άρα ήμασταν πιο έτοιμοι με το EFSF για να ξεκινήσουμε. Όπως είπε ο αξιότιμος κύριος στην τελευταία του ερώτηση, το πιο σημαντικό ήταν το εξής. Όταν αποφασίσαμε Μάιο 2010 εν το μέσο της νυκτός πράγματι πριν ανοίξει το χρηματιστήριο του Τόκιο έγιναν πολλά σωστά κάποια έγιναν κατά προσέγγιση και τότε τι αντιληφθήκαμε εκ των υστέρων ότι 440 δισεκατομμύρια δεσμεύτηκαν για το EFSF αλλά για να προστατεύσουμε το τριπλό α των μέσων έπρεπε να έχουμε κάποιο αποθεματικό το οποίο de facto μείωνε κατά το ίμιση περίπου τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Το ΙΦΣΕΦ από αυτό επηρεάστηκε. Και η όροι για τα επιτόκια επίσης. Για τη χώρα που έπαιρνε το δάνειο ήταν υψηλά. Εκ των υστέρων αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν η καλύτερη ρύθμιση και άλλαξαν εκ των υστέρων οι συνθήκες και οι όροι. Το FSF λοιπόν ένα ήταν πολύ πιο δαπανηρό από το EFSM για να βοηθήσουμε τις χώρες αποτελεσματικά το Συμβούλιο αποφάσισε τότε να κάνει το μοίρασμα που βάρινε περισσότερο το EFSM από ότι το EFSF. Μετά οι συνθήκες του EFSF 2 και το EFSM άλλαξαν για να γίνουν οι όροι λιγότερο επαχθείς για τις χώρες που έπαιρναν δάνειο. να επενθυμίσουμε ότι ναι μεν το EFSM έχει 60 δις η ανάληψη υποχρεώσεων του ESM για τις δύο χώρες Ιρλανδία και Πορτογαλία είναι λιγότερο από 36 δισεκατομμύρια και δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για περαιτέρω χρήση του EFSM μετά από τον Ιούλιο του 2012 όταν θα πάρει τη σκητάλη το ESM. Να θυμίσω και κάτι άλλο αφού μιλάμε για την έκθεση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσης ότι το ισοζύγιο το μέσο για το ισοζύγιο πληρωμών έχει 50 δις. Αυτά κατά τη διάρκεια της κρίσης διπλασιάστηκαν στα 50 δις και 11,4 δις έχουν δεσμευτεί. Άρθρο 122. Αυτή είναι η νομική βάση για την ίδρυση του FSM και διαβάζω από τη συνθήκη. Παράγραφος 2. Άρθρο 122. Λέει ότι όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή απειλείται σοβαρά με σοβαρές δυσκολίες που δημιουργούνται από φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικές περιστάσεις εκτός ελέγχου αυτού, το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να χορηγήσει υπό κάποιους όρους χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης στον λόγο κράτος μέλος ο πρόεδρος του Συμβουλίου θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ληφθήσεις αποφάσεις. Αυτή είναι η νομική βάση. Το άρθρο 122 που αναφέρεται σαφώς στο ρόλο του Κοινοβουλίου και πρέπει να πω ότι η νομική βάση για το EFSM επελέγει μετά από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κατεπίγουσα βοήθεια δυνάμει το άρθρο 122, ξεπερνώντας μια πολύ περιοριστική ερμηνεία όσον αφορά το άρθρο αυτό που αρχικά περιοριζόταν σε αυτά που σας διάβασα. Φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος μπορεί να προσθέσει κάτι από πλευράς του FSM. Θα ήθελα να σχολιάσετε το που Μάρκο Μπούτι για το διαμερισμό μεταξύ EFSF ή FSM. E Πέρα από το κόστος υπάρχει κάτι άλλο. Στην αρχή το e FSF ε, θεωρείται ο προσωρινός μηχανισμός και έτσι δημιουργήθηκε. Και υπήρχαν νομικέ απαιτήσει κυρίως πλευρά ενό κράτου μέλους, σύμφωνα με τις οποίε το FSF e θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί όταν απαιτείται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί άλλοι πόροι και υπήρξε σαφής λόγος να χρησιμοποιηθεί το EFSM εν πρώτης και μετά λιγότερα ποσά να βγουν από το EFSF. Ήταν πολιτική η προσέγγιση, πέρα από αυτά που ανέφερε ο Μάρκο Μπούτι. Θα ήθελα να πω όσον αφορά την προσωρινή ύπαρξη του, το EFSF δεν θα σταματήσει να υφίσταται, το 2013, τώρα το 2012 μάλλον, θα πρέπει να επομιστεί τις ευθύνες που πρέπει να διαχειριστεί. Από τη στιγμή που εκκρεμούν ομόλογα δάνεια θα εξακολουθεί να εφίσταται για τον έλεγχο της κοιτάλης του συνάδελφου από δεξιά. Ναι, να απαντήσω στην ερώτηση όσον αφορά τη τεχνική εξήγηση. Γιατί το FSF εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι τότε, το 2010, γι' αυτό. Πρώτον, πρακτική. Το FSF έπρεπε να είναι πολύ ευέλικτο. Οπότε η υποστήριξη θα χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το FSF είχε πολύ μικρό προσωπικό, λογιστικά, ταμείο, λογισμικό ανετίθετο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Αυτό ήταν ο πιο γρήγορο τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει, να βοηθηθεί να λειτουργεί το FSF. Είμαστε ακόμα σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και το EFSM, οι τραπεζικές δραστηριότητες, οι οικονομικές δραστηριότητες είναι στο Λουξεμβούργο. Άρα λογικό ήταν η ομάδα του Τόμας Γεράσιμος που είναι εκεί ε, να κινείται στο Λουξεμβούργο για να υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Και τα κράτη-μέλη ε, θεώρησαν ότι είναι λογικό να εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Για λόγους επιχειρησιακούς ήταν υποφελές να είμαστε στο Λουξεμβούργο. Δεύτερο ερώτημα για την PricewaterhouseCooper. Εδώ και δύο χρόνια πράγματι θεωρούνται σαν ο θεσμικός μας έλεγκτης και αυτή την ε, δράση ασκούν από την αρχή ύπαρξης του EFSF. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, θα ζητήσω να είναι πολύ σύντομη στο δεύτερο γύρο, συνάδελφοι. Άντρεάσεν, η κυρία Άντρεάσεν έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις. Μία, η πρώτη. EFSM. Σε περίπτωση χρεοκοπίας, Χρειάζεται να ζητηθούν συνεισφορές από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη δίνουν τα χρήματα για τα 60 δις και όχι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε. Δεν θα έπρεπε να προσβλέπουμε προς τα κράτη-μέλη και τι δυνατότητα έχουν να χρηματοδοτήσουν τη χρεοκοπία, εάν συμβεί μια χρεοκοπία. Δεύτερον, το EFSF γιατί εξακολουθεί να διανοδοτεί μετά τον Ιούλιο 2010 αφού θα υπάρχει ήδη το ESM. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Είπατε ότι το, το Συμβούλιο των Διευθυντών είναι ίδιο και το ίδιο προσωπικό. Έχει και τους ίδιους ελεγκτές. Τρίτον. Ποιος είναι υπεύθυνο για τη διαπραγμάτευση όρων για την εφαρμογή πολιτικών στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρομαι. Όταν υπέβαλε το πρώτο ερώτημα, απάντηση ήταν ότι θα ελέγχει συμμόρφωση. Η διαπραγμάτευση όρων για διαμόρφωση πολιτική είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Άρα, ερώτηση που απορρέει, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα έχει κάποια επιρροή όσον αφορά την διαπραγμάτευση για του όρου διαμόρφωση πολιτική. Ευχαριστώ, κύριε Άνδρασεν. Επόμενο, ο Γιάννη. Κύριε Πρόεδρε, έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα τις ε, συντομεύσω, τις πω περιληπτικά. Η πρώτη αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων στον κύριο Άνιβ. Όσον αφορά τη διευκρίνηση αυτής της σύγκρουσης συμφερόντων, προσανατολίζεστε σε διεθνείς προδιαγραφές, στον ε, ή έχετε κάποια άλλη αντίληψη για το πώς διευκρινίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και τι είδους μηχανισμοί επίλυσης προβλέπονται. Η δική μου εμπειρία είναι ότι όταν κάποιος από τις ε, χώρες ε, ε, όταν ε, διαπιστώνουν κάποιες αδυναμίες σε μια από τις χώρες ε, μέλη τελικά βγαίνουν τα μαχαίρια και δεν υπάρχει κάποια λύση. Το δεύτερο ερώτημα αφορά όλα τα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα στον κύριο Μπούτη. Ποιος καλύπτει τα διοικητικά έξοδα για αυτό το θεσμικό όργανο, ποια, σε ποιο ύψος εκτιμώνται και αν είναι η Κομισιόν αυτή που τα καλύπτει, κύριε Μπούτη, θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι στο πλαίσιο των επιπρόσθετων καθηκόντων που θα πρέπει να αναλάβει η Κομισιόν για αυτές τις λειτουργίες τότε ε, θα πρέπει να αυξηθούν, ε, θα αυξηθούν οι διοικητικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο ερώτημά μου απευθύνεται επίσης προ τον κύριο Μπούτη. Κάπω με εντυπωσιάζετε με την αισιοδοξία σας όσον αφορά τον αυτοματισμό της ε, αποπληρωμής εκ μέρου των χωρών μελών. Όλοι εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού γνωρίζουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά τις στάση των χωρών μελών όταν υπάρχουν δυσκολίες με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν, για παράδειγμα, ε, υπήρχαν μόνο τέσσερα δις ε, στα ταμεία πριν από μερικά χρόνια και έπρεπε να δοθούν 40 δις για, γεωργικές, ε, για πληρωμές στη Γεωργία. Άρα πώς μπορεί να αμβληθεί με τις συνεισφορές των χωρών μελών αυτός ο κίνδυνος για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν με πείσατε με την αισιοδοξία σας κύριε Μπούτη. Και ως τελευταία παρατήρηση θα ήθελα να πω το εξής. Το άρθρο 2 του ελέγχου του προπολογισμού ε, διατυπώνει κάποιες ε, συστάσεις για το EFSM Το ερώτημα έχει ως εξής. Σε ποιο χρονικό διάστημα θα απαντήσει η Κομισιόν αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάιερ. Ο συνάδελφος κύριο Ουντή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, εάν κατάλαβα καλά, να ρωτήσω το εξή. Τα 60 δις θεσμεύονται από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είναι μια, ένα εγγυητικό ποσό. Τι γίνεται στην αγορά των εγγυήσεων, αυτό αξίζει μεταξύ 0,3 ή 0,5%. Ε, οι δικαιούχοι αυτών των εγγυήσεων θα μας ανταμείψουν για αυτή την δέσμευση εγώ προσωπικά με το γεγονό ότι οι οίκοι αξιολόγηση τη πιστοληπτική ικανότητα επιτρέπουν ο πενιχρό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προσφέρει μία εγγύηση. Δεύτερον, η Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρεσίε τη αντιτίθενται στο η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να μπορεί να λειτουργεί ρυθμιστικά μεταξύ των ε, διαφόρων διακυβερνητικών θεσμικών οργάνων που έχουμε συστήσει, ούτω ώστε να διαφυλαχθεί η οικονομική σταθερότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα αυτή την πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους νομικής βάσης αντιτάχθηκε. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε γιατί αντιτάχθηκε η Επιτροπή και κατά πόσο αυτό είναι δικαιολογημένο και είναι δικαιολογημένο προτίθεται να κάνει μια πρόταση ούτω ώστε να έχουμε επιτέλους ένα ε, υπερεθνικό εργαλείο παρακολούθησης και τραπεζικής ρύθμισης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω η Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών εδώ και τέσσερα χρόνια ζητά ε, αυτή τη ρύθμιση της Διεθνούς Τράπεζας ε, Επενδύσεων η οποία στην περίπτωση αυτή θα χάσει το τριπλό α Έχουμε λοιπόν αυτή την ε, αρχή ε, η οποία έχει αυτή την αρμοδιότητα, αλλά η Επιτροπή αντιτάσσεται, αρνείται. Δεύτερον, θεωρείται να διευρύνει τις αρμοδιότητες αυτής της αρχής ε, επί τη βάση μιας συμπληρωματικής νομικής βάσης. Ευχαριστούμε κύριε Όντι. Αυτές ήταν κάπως μακρές, μακροτενείς ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ οι απαντήσεις να είναι σύντομες Επιτρέψατε μου να αναφερθώ εντάχει στο θέμα της συνεχής, συνεχής χρήσης του EFSF. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τα όσα είπε ο κ. Μπούτη και σχέση με τα όσα είπα ε, προηγουμένως για τις αποφάσεις του Eurogroup. Και αυτό σχετίζεται με την ε, τρέχουσα οικονομική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζομαι και τις απόψεις που υπάρχουν ε, μεταξύ των πολιτικά ηθινόντων και των αγορών ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα επαρκές τείχος προστασίας. Θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί το EFSF ενώ παράλληλα δημιουργούμε το τείχος προστασίας του ESM ε, χωρίς να προσθέτουμε αναγκαία σε αυτό για τα υπάρχοντα προγράμματα είναι 500 συν 200 το τείχος προστασίας τα οποία χρησιμοποίησαμε για την εξυπηρέτηση του ελληνικού δανείου πριν από το FSM. Νομίζω ότι η κινητήρια δύναμη εδώ ε, είναι το εφιστάμενο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το δεύτερο θέμα για την αιρεσιμότητα θεωρώ ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν μέχρι στιγμής. Δηλαδή ότι η αιρεσιμότητα θα συνεχίσει να επιβάλλεται, οι πολιτικοί όροι θα συνεχίσουν να διατυπώνονται όπως έγινε με το EFSF και για το ESM και αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στην έκθεση του PwC θα πρέπει να είναι συμβατό με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων που περιλαμβάνουν σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως μπορώ να ε, ξεκινήσω με το ESM όπως το EBRD και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να καλύπτει το δικό του κόστος. Θα έχει κέρδη και ζημίες, δηλαδή θα έχει ορισμένα έσοδα και στη βάση αυτών των εσόδων θα καλύπτεται το κόστος. Δεν θα είναι ένας κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά ε, και όπως οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα έχει τους δικούς του ανεξάρτητους λογαριασμούς για τα κέρδη και τις ζημίες. Όσον αφορά τις σύγκρουση ε, συμφερόντων, το ESM και στις λεπτομερείς διατάξεις του ε, ακολουθούνται οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Δηλαδή οι δικηγόροι και χώρες μέλη ε, βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στην περίπτωση σύγκρουσης ε, συμφερόντων των μελών και εξωματούχων αυτού του οργανισμού, αυτών των οργανισμών. Τώρα, όσον αφορά τον έλεγχο, κατά πόσο θα έχουν τους ίδιους ελεγχτές, το EFSF και το ESM, η δομή έτσι όπως την παρουσίαζα είναι κάπως διαφορετική. Το EFSF ε, θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία, θα έχει ελεγκτές που θα είναι ιδιώτη. στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι η PwC ή άλλοι ανταγωνιστέ του. για το ESM θα είναι διαφορετική η δομή θα υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο με πέντε μέλη και θα υπάρχουν νέοι ε, λογιστές οι οποίοι θα επιλεγούν ε, κάποιε κάποιες εταιρείες που θα κερδίσουν τον, ε, τον διαγωνισμό άρα δεν θα είναι οι ίδιοι ελεγκτές διότι πρόκειται για δύο διαφορετικές δομές αυτή θα είναι η προσέγγιση και αυτό θα γίνει μόνο εφόσον συσταθεί το ESM ε, την 1η Ιουλίου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Άνεφ. Ο κύριος Μπούτ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τέθηκαν πολλές ε, σημαντικές συζητήσεις που δίνουν πλούσια ρεθίσματα. Τώρα θα ήθελα να απαντήσω ορισμένες από αυτές. Καταρχήν το κατά πόσο οι ζημίες για τις ε, χώρες ε, μέλη και τον προϋπολογισμό τι γίνεται. Ε, προφανώς είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει κάποια προσημόμενη ποσά τα οποία συνδέονται με αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διάθεσή του στην περίπτωση ανάγκης και στην περίπτωση που οι χώρες μέλη είναι υποχρωμένες να συνεισφέρουν οι ίδιες είναι πολύ ξεκάθαρο όπως είπα προηγουμένως ότι η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το δικό της ταμείο εφόσον συντρέχει από χρόνο λόγος ε, και κατεξαίρεση. Και υπάρχει μια ειδική διάταξη του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισμού 1150 του 2000 που υποχρεώνει τις χώρες μέλη να ανταποκριθούν στο αίτημα της Επιτροπής και όπως αναφέρεται υπάρχει κάποιος ε, χρόνος, ε, μια προθεσμία 14 ημερών για το FSM να ε, την αιγίδα του FSM για τις χώρες μέλη και το πρόγραμμα στην περίπτωση της πληρωμής, πληρωμής εάν υπάρχει μια έγκαιρη, έγκαιρη προειδοποίηση ότι δεν έχουν φτάσει αυτές οι πληρωμές, τότε θα ενεργοποιήσουμε αυτές τις διατάξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 12. Και στην περίπτωση αυτή είναι μια υποχρέωση των χωρών μελών να το τηρήσουν, να συμμορφωθούν. Δεύτερο σημείο, όσον αφορά το κόστος διαχείρισης για την Επιτροπή. Όπως είπα, υπέρξαμε ιδιαίτερως ε, προσεκτικοί όσον αφορά την ευθυγράμμιση των όρων υπό το EFSM, για το EFSM ε, και για το EFSM και για το ESM. Άρα λοιπόν η αιρεσιμότητα είναι η ιδία για όλα τα όργανα, για όλα τα εργαλεία. Ε, εφαρμόζεται λοιπόν σε κάποιο πρόγραμμα και τα διάφορα εργαλεία παρέχουν τη χρηματοδότηση. Άρα το κόστος το οποίο συνδέεται με την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων έχει ενσωματωθεί στην κανονική παρακολούθηση αυτών των, τήρηση αυτών των όρων. Τώρα όσον αφορά τη δέσμη των 6 μέτρων, η αιρεσιμότητα αυτή είναι πιο αποτελεσματική, πιο αυστηρή ε, και είναι αυστηρότερη από ό,τι στο παρελθόν και αυτό ακριβώς γίνεται για να εξασφαλίσουμε τα προγράμματα εφαρμόζονται με έναν πλήρη τρόπο και υπάρχει μια πρόληψη του ώστε οι χώρες μέλη να μην ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα ε, ήδη στην πρώτη φάση. Όπως σας είπα προηγουμένως, μεταξύ του πακέτου των δύο και του ειδικού ευρωπαϊκού κανονισμού του Συμβουλίου που συζητιέται τώρα σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάναμε ακόμα πιο αυστηρούς τους όρους και επίσης θα υπάρξει μια παρακολούθηση μετά την εφαρμογή του προγράμματος, δηλαδή μια περίοδο που κανείς θα μπορούσε ενδεχομένω να θεωρεί ότι αν δεν υπάρχει μια τέτοια αυστηρή παρακολούθηση θα μπορούσε ενδεχομένω να επέλθει κάποια χαλάρωση όσον αφορά την εφαρμογή, την τήρηση των όρων. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει πιο αυστηρή την πολιτική αυτή της, των όρων ε, της, ε, της των 6 μέτρων ε, η οποία σε αυτή τη δέσμη των 2 μέτρων όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τώρα, όσον αφορά το προβληματισμό της ευρωπαϊκή Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αξιολογείται από τους οίκους ε, αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που βασίζονται στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 27 χώρες μέλη και είναι επαρκή η προστασία αυτή και θα ήθελα επίση να τονίσω τη συντηρητική διαχείριση του προπολογισμού. και ιδιαίτερος είναι αυτό το τελευταίο στοιχείο το οποίο στηρίζει ακριβώς το τριπλό α της, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης επίσης δίνουν ε, προσοχή στα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αυτό το οποίο προβλέπεται για το IFSF ε, κατοχυρώνει το τριπλό α για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνέχιση του τριπλού α. Τώρα, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κάποια διασύνδεση με τα εργαλεία διάσωσης, τα οποία δεν είναι τράπεζες, ε, αλλά δεν εφαρμόζονται σε αυτά. Παρ' όλα αυτά θα αποδώσουμε ένα ρόλο στην Ευρωπαϊκή τραπεζικέ αρχέ αρχές για ορισμένα εργαλεία, δηλαδή δικότερα στην περίπτωση της διευρυμένης δυνατότητας υποστήριξης υπό το EFSF και το ESM για δάνεια προς χώρες μέλη για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τόσο έντονη συζήτηση. Είδαμε τη, τα πράγματα από την προ, οπτική γωνία των όσων διαχειρίζονται τους τρεις μηχανισμούς και τώρα νομίζω Ήρθε η ώρα να ακούσουμε την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου. Όχι ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα ζητήματα, αλλά έχουμε εξαντλήσει σχεδόν το χρόνο μας. Άρα θα χρειαστεί να συνεχίσουμε σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχων των Προϋπολογισμών. Τώρα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ελεγκτικό συνέδριο. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Καλντέιρα και προτείνω να αρχίσετε αμέσως. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότυπο μέλη της Επιτροπής αξιότιμη, προσκεκλημένη. θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την κυρία Ιβανόβα για τη διοργάνωση ε, της ακρόας αυτής που θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στο ελεγκτικό συνέδριο μέσω εμού να ε, συμβάλλει στη συζήτηση. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής σας για τη διοργάνωση της ακρόας σχετικά με τους στόχους, τη λειτουργία και την ανασκόπηση ε, των μηχανισμών οικονομικής βοήθειας που συστάθηκαν ε, για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα ε, κρίση ε, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από το ελεγκτικό συνέδριο διότι συνιστά εξαιρετική ευκαιρία για μεγαλύτερη συνειδητοποίηση όλων των ζητημάτων που τίθενται όπως έχουμε δει σε προηγούμενες συζητήσεις Επίσης μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε παρελθούσες εμπειρίες ε, καθώς, όπου είναι και πιο σημαντικό, να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν. Ενδεχομένως στην παρουσίασή μου να υποπέσω στο λάθος της επικάλυψης, ε, της επακάλυψης, ε, ζητώ συγγνώμη. Αλλά είναι και καθησυχαστικό γιατί σημαίνει ότι έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση με τους λοιπούς προσκεκλημένους. Θα θυμάστε ότι εξ αρχής ήδη το 2010 ανέφερε με σαφήνεια το ελεγκτικό συνέδριο πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της πρέπει να ρίξει ιδιαίτερη έμφαση ε, στην ε, συμμόρφωση με βασικές αρχές πρέπει να διέπουν οποιαδήποτε χρήση δημοσίων κονδυλίων τον Νοέμβριο του 2010 παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Φαν Ρόμπεϊ, ε, το διευκρινίσαμε το ίδιο και σε ένα έγγραφο εργασίας που δημοσιεύσαμε το 2011 αναφερθήκαμε σε αυτή τη βασική αρχή. Πέραν αυτού το, τον Οκτώβριο του 2011, ε, σε συνεργασία με τις ανώτατες ελεγκτικές αρχές ε, των κρατών μελών στην ετήσια σύσκεψη που διοργανώνουμε στο ελεγκτικό συνέδριο επαναλάβαμε το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης. Νομίζω ότι αξίζει να το υπενθυμίζουμε, να υπενθυμίζουμε αυτές τις τρεις αρχές. Είναι πολύ απλές. Διαφάνεια, λόγοδοσία και δημόσιος έλεγχος. Διαφάνεια πρώτα απ' όλα Χρειαζόμαστε ε, αξιόπιστη και εμπρόθεσμη εγκαιρή ενημέρωση σε σχέση με την χρήση του ε, δημοσίου χρήματος ε, και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Στη συνέχεια, δημόσιος έλεγχος ούτω ώστε αυτοί που διαχειρίζονται τα προγράμματα και αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις να υπάγονται σε έναν έλεγχο. Ο δημόσιος έλεγχος είναι απαραίτητος σχετικά με την χρήση του δημοσίου χρήματος και τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται το δημόσιο χρήμα. Ε, ως προς αυτές τις τρεις βασικές ε, αρχές ε, εμπλέκεται το ελεγκτικό συνέδριο στη λειτουργία και των τριών μηχανισμών που αποτελούν και το αντικείμενο της σημερινής ακρόασης. Από τη δική μας οπτική γωνία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις ελέγχου του ελεγκτικού συνέδριου μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες, τρία διαφορετικά είδη ε, εργαλείων, αν θέλετε. Υπάρχουν ομοιότητες και βασικές διαφορές, όπως είπαν και οι προλαλείς. Θα αρχίσω με το EFSM και ε, το Μηχανισμό Βοήθειας ε, του Ισοζυγίου Πληρωμών, το BOP. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά θα υπενθυμίσω ότι βάσει τη συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται συγγνώμη, σαφή αρμοδιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την διαχείριση των κονδυλίων τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με αυτές τις συναλλαγές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε δανειοδοτική, δανειοληπτική ε, δραστηριότητα ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καταλογίζεται στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Οπότε υπάρχει πλήρες ελεγκτικό δικαίωμα ε, για το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της διαδικασίας χορήγησης δήλωση πιστείας από πλευρά του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Από το 2008 και μετά, όταν έχει να λειτουργεί ο μηχανισμό ε, ισοζυγίου ε, πληρωμών και ανήλθε στα 50 δις, με αποδέκτες κάποιες χώρες εκτός Ευρωζώνης, τότε είναι που ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2011. Επίσης, ενεργοποιήθηκε και τώρα επεξεργαζόμαστε τη διαδικασία χορήγησης δήλωσης αξιοπιστίας. Ελέγχουμε την ποιότητα της οικονομικής διαχείρισης δημοσιεύοντας ειδικέ εκθέσεις. Το Φεβρουάριο, αν θυμάστε καλά, συζητήσαμε μια τέτοια και θα αρχίσουμε τώρα τον έλεγχο των συστημάτων ισοζυγίου πληρωμών και του EFSM. Το δεύτερο είδος εργαλείων είναι η ο μηχανισμός για τα ελληνικά δάνεια, Greek Loan Facility, εδώ δεν απορρέουν από τη συνθήκη, τουλάχιστον άμεσα, οι αρμοδιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου Δεν εμπλέκεται δηλαδή αυτός κάθε αυτός ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Στην πράξη όμως έχουμε ρυθμίσεις για διακρατική συνεργασία και ο κίνδυνος βαρύνει κυρίως τα ε, εθνικά ταμεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει τον εξή ε, βασικό ρόλο να προσδιορίζει ε, τη, τα κριτήρια συμμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στην εποπτική διαδικασία και Βάσει πάλι τη συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωση ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο τι διοικητικέ δαπάνε όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών ε, οργάνων ε, καθώς ε, και την λειτουργική αποδοτικότητα τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ελέγχουμε λοιπόν τη διαχείριση από πλευρά αυτών των θεσμικών οργάνων. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στην Επιτροπή σα ότι είναι περιορισμένη η πόρη μα και άρα οφείλουμε να ιεραρχούμε προτεραιότητές μας ως προς την ελεκτική μας δραστηριότητα και να τις μοιράζουμε ανάμεσα ε, στον προϋπολογισμό και στα επιμέρους ε, προγράμματα χρησιμοποιώντας ε, μία σειρά από διαφορετικά κριτήρια αξιοποιώντας το έπακρο τους περιορισμένους μας πόρους. Τέλος, ESM, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο πιο νέος από όλους που θα διαδεχθεί μόνιμα τους ε, προσωρινούς μηχανισμούς EFSF και FSM. Ε, ως προς την μετάβαση από τους δύο αυτούς μηχανισμούς στον μόνιμο μηχανισμό, οφείλουμε να αναρωτηθούμε ε, πώς ακριβώς θα γίνει και οι μεταβατικές διατάξεις δεν έχουν πλήρως ε, προσδιοριστεί για το EFSF. Ε, ε, πήραμε κάποιες πληροφορίες από τον κύριο Άνε, θα ακούσουμε και το γερμανικό ελεγκτικό συνέδριο στη συνέχεια, αλλά για το EFSM ε, ήθελα να σας πω ότι, για το ESM μάλλον, είναι σαφές ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα να ελέγχουμε αυτόν τον μηχανισμό, αυτήν την νομική οντότητα. Αυτό είναι σαφές. Όπω ακούσαμε και στην παρουσίαση του κυρίου Άνεφ, έχουμε το δικαίωμα να διορίζουμε ένα από τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ESM. Αυτό συνιστά με ε, σοβαρή προσθήκη σε όλες ε, τις ε, διατάξεις που προβλέπονται στην συνθήκη σύστασης του ESM. Δεν ε, θα υψέλθω σε λεπτομέρειε για τη σύνθεση αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι θα μα απασχολεί στη συνέχεια. Αφήστε που το περιέγραψαν και οι προλαλήσαντε, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι όπως και στο EFSF η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαδραματίσει κέριο ρόλο για την προετοιμασία και την λειτουργία των εθνικών προγραμμάτων αναπροσαρμογής. θα έχουμε μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης, ανάλυσης και διαχείρισης ακινδύνου παραδείγματος χάρη και ε, θα πρέπει εμείς να υποπτεύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν είναι πρόσφορο να διαδραματίζει η Επιτροπή ε, το ρόλο αυτό στα πλαίσια του ESM. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί που εξετάζεται σήμερα εντάσσονται σε μια ευρύτερη ε, ανταπόκριση, αν θέλετε, από πλευράς πολιτικής με στόχο να αναβαθμιστεί η οικονομική διακυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, παραδείγματο χάρη. Πέρυσι μας απασχόλησε ιδιαίτερος. Έχουμε την δέσμη των έξι οδηγιών και ε, πρόσφατα είχαμε και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Επίσης, ο κανονισμός για τη μεταρρύθμιση και την εποπτεία των αγορών που μας οδήγησε στην ε, ίδρυση τριών νέων εποπτικών αρχών όπου φέρει την ευθύνη ελέγχου ε, πάλι το ελεγκτικό συνέδριο. Εφόσον είναι ιδιαίτερα ε, σημαντική η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων, τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο μελέτης ε, με στόχο ε, προσαρμογή της διαδικασίας, ούτω ώστε να έχουμε πιο αξιόπιστες ε, στατιστικές ε, πληροφορίες. Σε σχέση με τις ευθύνε και τις υποχρεώσεις του, το ελεγκτικό συνέδριο οφείλει να χρησιμοποιήσει τη μοναδική θέση και προοπτική που διαθέτει, ούτω ώστε να βελτιώνει την λόγοδοσία, την διαφάνεια και τον δημόσιο έλεγχο κατά την εφαρμογή αυτών των αρχών, συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα συμβάλλουμε ανα περίσταση, όχι μόνο ως αντίδραση για την τρέχουσα κρίση, αλλά και ως προς την αποτίμηση του γενικότερου ευρωπαϊκού τοπίου, με άξονες πάλι το δημόσιο έλεγχο, την λογοδοσία και τη διαφάνεια. Για να επανέλθω στο ESM, οι διατάξεις περί εξωτερικού ελέγχου είναι πολλά υποσχόμενες, ε, χάρη και στο διακυβερνητικό χαρακτήρα αυτού του μηχανισμού, κυρίως αν κάνουμε μια παραβολή με τον προκάτοχο, το EFSF. Ο λόγος ύπαρξης του ESM είναι να διαφυλάξει την ακαιρεότητα της Ευρωζώνης και άρα συνιστά ένα από τους βασικούς πυλώνες της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης που συνιστά με τη σειρά τη θεμελιώδη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτού κλείσω θα ήθελα να τονίσω, Πρόεδρε, ότι η συνεργασία ανάμεσα στις Εθνικές Ελεγκτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τελεσφόρησε μέχρι στιγμής. Έχουμε την ομάδα επαφής ε, που δραστηριοποιείται ε, στα πλαίσια της Ευρωζώνης ε, που μας επιτρέπει να προετοιμάζουμε κοινέ θέσεις οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αναθεωρημένη συνθήκη για το ESM και εσχάτως και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Στρέφομαι κυρίως προς τους Γερμανούς συναδέλφους που έχουν ηγετικό ρόλο ε, σε αυτόν τον τομέα. Το ε, αυτό στο οποίο πρέπει να αποσκοπούμε είναι καλύτερο συνδρομός, καλύτερη συνεργασία, ούτω ώστε να έχουμε καλύτερο δημόσιο έλεγχο, διαφάνεια και λογοδοσία, διότι αυτές είναι βασικές προτεραιότητες ε, και νομίζω ότι τονίστηκε παρκώς στη σημερινή ακρόαση. Τέλος. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, έχουμε αναλάβει δέσμευση να σας ε, υποστηρίζουμε να σας συνδράμουμε κάθε φορά που υπάρχει χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού της Ένωσης με στόχο πάντοτε τον καλύτερο δημόσιο έλεγχο, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ευχαριστούμε κύριε Καλντέιρα όχι μόνο για αυτά τα πολύτιμα εισαγωγικά σχόλια που κάνατε ε, σε σχέση με τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά καθώς και για την έμφαση που αποδώσατε σε αυτές τις αρχές της διαφάνειας και του δημοσίου ελέγχου. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο των δυνατοτήτων ελέγχου και τις ε, ε, προκλήσεις από ευρωπαϊκή σκοπιά να περάσουμε στα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Horst Erb που είναι μέλος του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και επικεφαλής στο τμήμα της για τη συνεργασία με την Επιτροπή Προπολογισμού της Γερμανικής Βουλής και εκπροσωπεί τώρα τον Γερμανό Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Ιβάνοβα, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω μέρος σε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα επίσης να διαβιβάσω θερμούς χαιρετισμούς από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Έγγελς, ο οποίος επίσης ε, είπε ότι είναι ιδιαίτερος ευγνώμων το θέμα του εξωτερικού οικονομικού ελέγχου που σχετίζεται με τους ε, μηχανισμούς ε, διάσωσης μπορούν να παρουσιαστούν τα θέματα αυτά και από μια εθνική σκοπιά. Η συζήτηση μέχρι τώρα και οι παρουσιάσεις των εκπροσώπων της Επιτροπής και των μηχανισμών διάσωσης έδειξε ότι αυτά τα μέτρα υποστήριξης για το ευρώ δεν αφορούν μόνο ευρωπαϊκά χρήματα, δηλαδή χρήματα της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, αλλά σε μεγάλο βαθμό ε, και εθνικούς προϋπολογισμούς και υπάρχουν τεράστιες υποχρεώσεις εγγύησεων που βαρύνουν τις χώρες ε, μέλη και που θεμελιώνονται στις ε, συνθήκες αυτές. Και αυτό θέτει κατά ανάγκη το ερώτημα ποιος ελέγχει αυτά τα δημόσια κονδύλια από εθνική πλευρά στις χώρες μας, στην ε, Ευρώπη και αυτό είναι απολύτως αυτονόητο. Η χρήση δημοσίων πόρων ε, ελέγχεται από ανεξάρτητα ελεγκτικά συνέδρια τα οποία υποβάλλουν εκθέσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια για τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου και με τον τρόπο αυτό διενεργούν τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο με έναν αυτονόητο τρόπο που όσον αφορά τα δημόσια κονδύλια είναι απολύτως αναγκαία. Γι' αυτό ε, ε, λάβαμε μέλος σε μια διαβούλευση με το Γερμανικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του περασμένου έτους και για πρώτη φορά παρουσιάστηκε ένα σχέδιο της τελικής συνθήκης και διαπιστώσαμε ότι σε αυτή τη συνθήκη δεν προβλέπεται εντολή για έναν ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο. Δεν προβλέπεται λοιπόν μια τέτοια εντολή και η συνθήκη ναι μεν προβλέπει έναν εσωτερικό έλεγχο αλλά δεν περιλαμβάνονται κάποιες σκέψεις, κάποια πρόβλεψη για έναν εξωτερικό έλεγχο. Ωστόσο αυτό δεν συμφωνεί με τις, τους διεθνούς κανόνες ε, για, ε, που ισχύουν διεθνώς ε, για παράδειγμα το, τη διάταξη 5.000 που προβλέπει ότι θεσμικά όργανα τα οποία χρηματοδοτούνται από δημόσιους προπολογισμούς ε, υποβάλλονται ε, στον έλεγχο των ανώτατων ελεγκτικών εποπτικών οργάνων που δεν εξετάζουν μόνο τη χρήση των κονδυλίων και ζητήματα κανονικότητας αλλά και πτυχές οικονομικότητας οικονομικά ζητήματα και αυτό προβλέπεται για διεθνή θεσμικά όργανα και την υποχρέωση εξωτερικού ελέγχου. Και απευθύνθηκαμε λοιπόν στον Υπουργό Οικονομικών και παρουσιάσαμε το θέμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού στη Γερμανία και αυτό ελήφθη υπόψη και ο Υπουργός παρακάλεσε στη συνέχεια να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες ούτως ώστε ή δυνατόν ε, διάφορα ευρωπαϊκά ελεγκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλουν σχετικά κάποιες προτάσει για αυτό το έλλειμμα. Και στη συνέχεια ακολούθησε μια συνάντηση τον περασμένο Σεπτέμβριο που εκπρόσωποι των Εθνικών Ελεγκτικών Συνεδρίων και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συναντήθηκαν με τον εκπεφρασμένο στόχο πρωτίστως να υποβάλουν μια πρόταση για μια διατύπωση ε, πρόβλεψη εξωτερικού οικονομικού ελέγχου που περιληφθεί στην τελική συνθήκη, δηλαδή πώς φαντάζονται αυτόν τον εξωτερικό έλεγχο και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συνθήκη. Δεύτερον, ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση χρόνου, γιατί η συνθήκη ήδη, το πρώτο σχέδιο μάλλον της συνθήκης είχε ήδη υπογραφεί. Άρα λοιπόν, τι είδου διαβήματα ήταν αναγκαία, ούτω ώστε να συμπεριληφθεί αυτή η διάταξη στη συνθήκη. Και τότε τα ελεγκτικά συνέδρια στη συνέχεια... Ε, ε, διατύπωσαν μια τέτοια ρύθμιση περιλαμβάνει έξι σημεία. Πρώτον, δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου με έξι μέλη, ε, ανώτατες ελεγκτικές αρχές των χωρών μελών. Αυτή ήταν η βασική αφετηρία. Και το Συμβούλιο αυτό, το ελεγκτικό αυτό Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει εποπτικό ρόλο έναντι των εσωτερικών ελεγκτικών οργάνων και θα έπρεπε ε, πέρα από αυτό να εξετάζει τους οικονομικούς κινδύνους και την ε, διαχείριση του προγράμματος και επίσης να είναι αρμόδιο ε, να υποβάλει εκθέσεις για τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτές οι πρωτοβουλίες των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων, όπως είπε ο κύριος Καλδέρο, αντανακλάται στην Επιτροπή Επαφών των Ανώτατων Εποπτικών Αρχών, Όλα δηλαδή τα Εθνικά Ελεγκτικά Συνέδρια, συνέδρια συγγνώμη, και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συζήτησαν και πήραν από αυτό το όργανο την Επιτροπή Επαφών, την πλήρη τους έγκριση. Ο, Καλδέρα, ο κ. Καλδέρα τότε απευθύνθηκε και στα Εθνικά Κοινοβούλια και, στο Ευρωπαϊκό, και στα Ευρωπαϊκά Όργανα για να υποβάλει αυτή την πρόταση. Εμείς στη Γερμανία αλλά και άλλα ελεγκτικά συνέδρια της Ευρωζώνης απευθύνθηκαμε και πάλι στα Εθνικά Κοινοβούλια και στα Υπουργεία Οικονομικών ε, ε, ζητήσαμε να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση για, ένα ε, για μια τέτοιου είδους ρύθμιση. Η πρωτοβουλία ήταν πετυχημένη κατά την άποψή μας και υπάρχει ένα άρθρο 30 εντωμεταξύ στη συνθήκη για το FSM και αυτό το άρθρο 30 αναφέρεται στους, ε, στα βασικά σημεία όσων είχαμε θέσει εμεί εκ μέρου των, των Εθνικών Ελεγκτικών Συνεδρίων και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό τη μορφή προτάσεων. Και στη συνέχεια ε, θα υπάρξει αυτή η ελεγκτική επιτροπή, έχει πέντε μέλη, δεν θα πρέπει να υπάρχουν όλοι από ελεγκτικά συνέδρια, αλλά τρία ναι ε, και δύο από εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και χαιρετίζουμε το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει μία μόνιμη εντολή και θα υπάρξουν και άλλοι εμπειρογνώμονες που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το εποπτικό όργανο, κάτι το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι χρήσιμο για την σωστή λειτουργία αυτού του οργάνου. Σημαντικό είναι τα μέλη να αναλάβουν προσωπικά την εντολή τους. Αυτό σημαίνει όσοι προέρχονται από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, όπως διορίζονται, θα πρέπει να αναλάβουν προσωπικά ε, δραστηριότητα ε, δεν είναι υπόλογα, αλλά είναι μια προσωπική εντολή. Δεν ε, δέχονται λοιπόν εντολές από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Επίσης, στη συνθήκη αναφέρονται συγκεκριμένα προσόντα για αυτά τα πρόσωπα και θα πρέπει να, είναι, ε, να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν κανονικά το έργο τους. Επίσης, ε, το Συμβούλιο Διοικητών υποβάλλει μία έκθεση και την διαβιβάζει στα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωζώνης επίσης στα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια ε, δεν πρόκειται για μια δεν υπάρχει μια ε, ειδική νομική ρύθμιση για το πώς θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαβίβαση, αλλά νομίζω ότι από τη συζήτηση που έγινε εδώ προέκυψε ξεκάθαρα ότι μια τέτοιου είδου έκθεση ασφαλώς θα πρέπει να βρει το δρόμο της και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, το άρθρο 30 λοιπόν είναι σημαντικό βήμα για τη συνθήκη του FSF όσον αφορά την εδραίωση του εξωτερικού ελέγχου, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν και άλλες ελλείψεις. Το Μάρτιο αυτού του έτους συναντηθήκαμε και πάλι στη Βόνη και ε, υποβάλαμε κάποιες ε, προτάσεις και ε, τις επεξεργαστήκαμε εν σχέση με το πώς μπορεί να γίνει αφενός μια διευκρίνηση των διατάξεων του άρθρου 30 και δεύτερον πώς ε, είναι δυνατόν να απαντηθούν κάποιες ε, εκκρεμείς ακόμα κατά την άποψή μας ερωτήσεις ε, μέσω των λεγόμενων bylaws, των λεπτομερών διατάξεων. Η πρότασή μας εδώ για τα bylaws, για τις λεπτομερείς διατάξεις, είναι να οριστεί επακριβώς ο χρόνος θητείας των μελών. Η πρότασή μας είναι τρία έτη. Τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να διορίζονται προσωπικά για τρία έτη. Δεν θα πρέπει να εμφανίζουν σύγκρουση συμφερόντων και επίσης ε, λέγεται κάποια πράγματα σχέση με το σύστημα της, ε, του εκπεριτροπής διορισμού αυτών των μελών και επίσης είπαμε ότι το Συμβούλιο αυτό θα πρέπει να κάνει κάποιο, ε, κάποιους ελέγχους για την οικονομική αποδοτικότητα και επίσης για το θέμα της διαχείρισης των κινδύνων για το EFSM που ε, Πέρα από αυτό, στι συστάσει που έχουν επεξεργαστεί εδώ, ε, συμπελήθησαν κάποια τεχνικά θέματα, για παράδειγμα το πώ τα μέλη των Επιτροπών μπορούν να προσφύγουν σε εμπειρογνώμονε. Επίση, ζητήθηκε να υπάρξει μια ρύθμιση η οποία να λέει το έργο του Συμβουλίου να υποστηρίζεται από το ESM Και επίση ζητήματα κόστου ε, τέθηκαν όσον αφορά τι απάνε ταξιδίου, τα έξοδα για του εμπειρογνώμονε κλπ. Όλα αυτά είναι προτάσει που κατά την άποψή μα ε, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στι λεπτομερεί διατάξει, τα bylaws. Και πλέον οι σχετικές προτάσεις έχουν φτάσει στα αρμόδια όργανα για τις λεπτομερεί διατάξεις, τα bylaws και ελπίζουμε ότι θα ληφθούν εκεί υπόψη. Υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Έρπ για, τα, για όσα μας είπατε και θα ήθελα να δώσω λόγω του προκεχωρημένου της ώρας το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Βαν Βάντεμπος από το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο γιατί εκπροσωπεί τον αντιπρόεδρο του Ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Βέντριξ, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Κύριε Βάνμπος, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Χαιρετίσματα στον κύριο Χέντριξ. Και περιμένουμε να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Περνάμε δύσκολους καιρούς, κυρίε και κύριοι. Χθε η κυβέρνησή μας έπεσε. Και το ίδιο βράδυ ε, αρρώστησε και ο βουλευτής μας. Και δυστυχώς δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα και ζητά συγγνώμη. Θα ήθελε πάρα πολύ να μιλήσει ο ίδιος προσωπικά εδώ σε αυτή την ακρόαση, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορεί. Μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους του και αυτό θα κάνω. Κυρίες και κύριοι, ανώτατοι ελεγκτικοί φορείς έχουν ευθύνη να προωθήσουν την ε, λογοδοσία και τη διαφάνεια σε δημόσιες στεριότητες που χρησιμοποιούνται δημόσιοι πόροι. Αυτό δεν είναι μόνη άποψη του δικού μας θεσμικού οργάνου, του Ολλανδικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά άποψη όλων των πλευρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρόσφατα σε ψηφίσματα ε, έχουμε αναφερθεί στο θέμα όσον αφορά την οικονομική κρίση. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και άλλα εργαλεία της σταθερότητας που έχουν δημιουργηθεί ε, μέσω αυτών λαμβάνουν άνευ ε, προηγουμένου, για άνευ ποσά Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσεις όχι μόνο από τα κράτη-μέλη της, Ευρωζώνης δεν λαμβάνονται αλλά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς χρηματοστηρικούς οργανισμούς για να πετύχουμε και να διατηρήσουμε δημόσια υποστήριξη για αυτά τα μέσα, διαφανής λογοδοσία για αυτά που αναλαμβάνονται και ε, να είναι υπόλογοι αυτοί που ασχολούνται ε, με τις λειτουργίες αυτές και καλή ανεξάρτητη έλεγχη είναι απαραίτητη. Σύμφωνα με το Ελεκτικό Συνέδριο της Ολλανδίας, το μέσο η σταθερότητα, τα μέσα που έχουν αναπτυχθεί, δεν αναπτύσσουν και δεν λαμβάνουν επαρκώ υπόψη αυτέ τι αρχέ. Η συμμόρφωση με αυτέ τι αρχέ θα πρέπει να ισχυθεί στο μόνιμο μηχανισμό που συστήνεται. Για να είμαι πιο ακριβή, πιστεύουμε ότι οι διευθετήσει των μέσων σταθερότητα ε, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τρει απαιτήσει. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή διαφάνεια υπό την μορφή αξιόπιστων και εγκαίρων πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων εθνικών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την παρούσα χρήση και την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι και τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται αυτοί οι δημόσιοι πόροι. Δεύτερον, χρειάζεται να υπάρχει επαρκή έλεγχο, λογοδοσία, να υπάρχει δημόσιο έλεγχο των επιχειρήσεων και θα πρέπει να είναι υπόλογοι εκείνοι που παίρνουν τι αποφάσει και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των διαφόρων διαδικασιών. Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή δημόσιο έλεγχο να παρέχονται διαβεβαιώσεις και πληροφορίες για τη χρήση των δημοσίων πόρων και των κινδύνων στον οποίο εκτίθενται. Έτσι θα συμβάλλουν στη διαφάνεια και θα παρέχεται μια βάση για, την, ε, τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Α εξετάσουμε από το σύνεγγυ στο ESM. Αυτό το εργαλείο για τη χρηματοσυντική σταθερότητα δημιουργήθηκε επί τη βάση διακυβερνητική συνθήκη που υπεγράφει από τα 17 κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη. Θα είναι ένα διεθνή οργανισμό ε, νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το δημόσιο, Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο. Όπως περιγράφεται στη μελέτη που διενεργήθηκε για την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών, οι ρόλοι και οι διευθετήσεις των διοικητικών φορέων της ESM καθορίζονται σαφώς και ευθυγραμμίζονται με την κοινή πρακτική που εφαρμόζεται από διεθνείς φορείς ε, παροχή σηματοστική ενίσχυση όπω το Δούνου του Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Το ESM όμω δεν ταιριάζει στην ε, νομική τάξη και το το θεσμικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, παρόλο που η τροποποίηση συνθήκη τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ήταν κάτι απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και κάποιοι, όπω το Εθνικό, το Ανώτατο Συμβούλιο τη Ολλανδία, στι γνωμοδοτήσει που επικύρωνε τη συνθήκη του ESM, τροποποιώντα το άρθρο 136 TFEU, ε, επιχειρηματολόγησε λέγοντα ότι αυτό ήταν μια σκόπιμη επιλογή. Οι ρόλοι και αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ενώση όσον αφορά το ESM είναι περιορισμένοι και σημαντικέ διατάξει όσον αφορά το δημοκρατικό και νομικό έλεγχο, δικαστικό έλεγχο δεν έχουν συμπεριληφθεί στη συνθήκη για το ESM. Ενώ μεν ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο ρόλο που θα παίξουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο ESM είναι κρίσιμο, η ανάλυση τη σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τη χρηματοδοτική σταθερότητα του ευρώ η διαπραγμάτευση του Μνημονίου Συνεννόησης με τα μέρη, ε, μέρη του ΕΣΕΜ που ζητούν οικονομική σταθερότητα, η λεπτομερή αιρεσιμότητα όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυση, η παρακολούθηση μόρφωση με την εφαρμογή τη αιρεσιμότητα, επαρκέ προβλέψεις για δημοκρατικό έλεγχο και αποτελεσματικό εξωτερικό έλεγχο όσον αφορά τα καθήκοντα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής λείπουν από τη συνθήκη του ΕΣΕΜ η μόνη άλλη αναφορά ρητή εκτός από το άρθρο 13 ε, όσον αφορά τα καθήκοντα βρίσκονται μόνο στο προήμιο όπου εκεί αναφέρεται ότι η εποπτεία μετά τα προγράμματα θα εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσης που καθορίζει τα άθρα 121 και 136. Ποιος θα φέρει την ευθύνη όμως για τον έλεγχο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμορφώθηκε τα καθήκοντά τη όσον αφορά το ESM. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο των Ελεκτικών Φορέων, η συνθήκη δίνει στο, στο Συμβούλιο των Ελεκτών συγκεκριμένο καθήκον όσον αφορά τον έλεγχο των λογαριασμών του ESM, σύμφωνα 30, και την επαλήθευση των λειτουργικών λογαριασμών και του σωζυγίου το, ναι, το Συμβούλιο των Ελεκτών μπορεί να διενεργεί ανεξαρτήτους ελέγχους και να έχει πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα του ESM που, αφαιτούνται που για την ε, λειτουργία του. Σύμφωνα με την Ολλανδική κυβέρνηση αυτές είναι απλώς οι βασικές διατάξεις και μπορούν να επεκταθούν μέσω των λεπτομερών διατάξεων εσωτερικού κανονισμού που συντάσσεται. Το... Κάτω, η κάτω βουλή της Ολλανδίας Υιοθέτησε δύο νομοσχέδια επί του θέματος και η Ολλανδική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί ούτω ώστε να εφαρμόζεται πλήρη εξωτερικό δημόσιο έλεγχο και να υπάρχει πλήρη ε, διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά την ε, χρήση των πόρων του ΕΣΕΜ. Όπως ανέφεραν μόλις τώρα οι Γερμανοί συνάδελφοι, θα ήθελαν οι διάφοροι φορεί σηματοψηφική ανθρωπή Ευρωπαϊκή Ενώσεω να δουν ότι το ελεκτικό αυτό συμβούλιο θα μπορεί να ελέγχει τακτικά συμμόρφωση, επιδόσει και διαχείριση κινδύνου πλευρά ESM. Και τώρα γίνονται συζητήσεις για τον εσωτερικό κανονισμό του, του ESM ε όταν ξεκίνησε να λειτουργεί και εμείς έχουμε εκφράσει επιθυμίε επιθυμίες με τη βοήθεια των κυβερνήσεών μας αυτές οι επιθυμίες ελπίζουμε να ληφθούν υπόψη και να υιοθετηθούν. Όμως αν αυτό δεν γίνει ίσως ο μόνος έλεγχος αποτελεσμάτων και συνεπιών των ε, λειτουργιών του ESM ε θα είναι ειδικές, ειδικοί έλεγχη από πλευρά ΙΚΑ ε, των δραστηριοτήτων που διενεργείται από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, βάσει των άρθρων 121 και 136. Οι διάφοροι ελεγκτικοί φορεί των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν έχουν ίδιο δικαίωμα να ελέγξουν ένα διεθνή οργανισμό. Ο πρωταρχικό στόχο του είναι να ελέγξουν τι εθνικέ κυβερνήσει και το πώ δαπανούν τα δημόσια χρήματα. Οπότε έτσι γίνεται δύσκολο για ελεκτικού φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώση να κάνουν περισσότερα από αυτά που κάνουμε του παρόντο μέσω τη ιστοσελίδα μα www.recordcamer.nl κάθετο EU Pavla Governance Pavla EN που δίνει πλήρη εικόνα όσον αφορά τις γρήγορα μεταλλασσόμενες εξελίξεις στον τομέα και έτσι βοηθά να δημιουργείται διαφάνεια για το Εθνικό Κοινοβούλιο και για το γενικότερο κοινό. Για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, η έλεγχη όσον αφορά τις συνέπειες και αποτελέσματα των λειτουργιών του ΕΣΕΜ είναι κάτι σχετικά καινούριο, διότι το καθήκον του ελέγχου, δηλαδή εξετάση του εισοδήματο και των δαπανών τη Ένωση, παραδοσιακά ερμηνευόταν περιοριστικά. Τέτοιοι έλεγχοι επιπλέον θα λαμβάνουν χώρα εκτό του πλαισίου ESM και μόνο είναι, θα είναι ένα έμεσο έλεγχο των ε, λειτουργιών του ESM. Από την έποψη του ιδίου του ESM, δεν, είναι, δεν αρκεί σαν δημόσιο έλεγχο του ESM αυτό. Α σκεφτούμε εν συντομία ποιε είναι οι δύο άλλε πτυχέ ε, τη διακυβέρνηση ESM που αναφέρονται. Η διαφάνεια δηλαδή και η λογοδοσία. Έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίε μεν για να ενισχυθεί η διακυβέρνηση του ESM όσον αφορά το δημόσιο έλεγχο. Οι διευθετήσει που διατυπώνονται στη συνθήκη ESM για διαφάνεια και λογοδοσία είναι ε, αδύναμε. Και από ό,τι γνωρίζουμε, τίποτα συγκεκριμένο πέρα από την ακρόαση που διεξάγεται σήμερα γίνεται για να αλλάξει αυτό. Σύμφωνα με τη συνθήκη για την ESM, η ESM θα δημοσιεύει ετήσια έκθεση που θα περιέχει δήλωση που θα έχει ελεγχθεί όσον αφορά τους λογαριασμούς της και θα υποβάλει στα μέλη του ESM ε, τρίμηνη δήλωση όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση, κέρδη, απώλειες όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Δυνάμει άρθρου 27. Το Συμβούλιο των ε, Ελεγκτών θα συντάσει ετήσια έκθεση επίσης για την υποβάση στο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι προσβάσιμη έκθεση αυτή στα Εθνικά Κοινοβούλια, του ελεγκτικούς φορείς των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ενώ ο περιορισμένος, το περιορισμένο πλαίσιο της αναφοράς ελέγχου που θα συστήνεται από το ESM δημιουργεί προβλήματα, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ολλανδίας πιστεύει ότι τίποτα δεν τίθεται δημόσια, ότι αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό. Χωρίς μοίρασμα πληροφοριών και έλεγχο του κοινού, πώς θα είναι δυνατόν να αποκτήσει κανεί και να διατηρήσει την υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών. Θα θέλαμε, παραδείγματο χάρη, να δούμε ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργείται από το Συμβούλιο των Ελεγκτών να διατίθεται στο διαδίκτυο. Στη γνωμοδότηση για τη συνθήκη του ESN, το Ανώτατο Συμβούλιο τη Ολλανδία ε, δηλώνει ότι η σημαντική συνέπεια τη επιλεχθήση διακυβερνητική δομή είναι ότι οι φορεί του ESM δεν είναι υπόλογε ε, στα πλαίσια τα θεσμικά τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως Επιπλέον αναφέρει ότι το ESM δεν έχει δικαστική ασυλία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παίζει κανένα ρόλο, το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν έχει δικαιώματα ελέγχου αυτό καθε αυτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να ασχοληθεί μόνο με διαφορές ε, ε, και προσφυγές κράτους, μάλλον μέρους του ESM. Δημοκρατικό έλεγχο και δημόσιο έλεγχο υπάρχει στον περιορισμένο βαθμό που οι Υπουργοί Οικονομικοί μπορεί να είναι υπόλογοι από πλευρά Εθνικών Κοινοβουλίων για το μερίδιο του ε, συμμετοχή στο ESM και όχι για τη λειτουργία του ESM και των φορέων του ESM ούτε του ίδιου του οργανισμού. Το ανώτατο συμβούλιο ε, της Ολλανδίας θεωρεί ότι ο ελληπής δημοκρατικός έλεγχος είναι κάτι προβληματικό κυρίως λόγω της ε, μόνιμης φύσεως του μηχανισμού σταθερότητα και του όγκου του οικονομικού. Ε, στην γνωμοδότησή του η, η παρούσα διακυβερνητική μορφή δεν μπορεί να είναι τελικό αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας της διαμόρφωσης οικονομικής διακυβέρνησης αλλά απλώ ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Η Ολλανδική κυβέρνηση όμως διαφωνεί. Η ε, ε, λογοδοσία που δίνει στο Εθνικό Κοινοβούλιο για το ESM ξεπερνά αυτά που δίνονται σε άλλους διεθνείς σηματοστικούς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ. Σύμφωνα με την Ολλανδική κυβέρνηση, αυτό σε συνδυασμό με την εμπλοκή των ελεκτικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου στη συνθήκη ESM οδήγησε σε μια επαρκή βάση, ότι εξασφαλίζεται ο δημόσιο δημοκρατικό έλεγχο του ESM. Ενώ το ελεκτικό συνέδριο το, της Ολλανδίας ε, χαιρετίζει τη δημοκρατική επιρροή από πλευρά της Ολλανδικής κυβερνήσης, που δίνεται την Ολλανδική κυβέρνηση, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εξέφασε το Ανώτατο Συμβούλιο της χώρας μας όσον αφορά ε, τον, την επικύρωση της συνθήκης ESM. Οι περιορισμοί που αφορούν τη διαφάνεια και την ε, λογοδοσία είναι μεγάλοι. Και αυτό με τις ανησυχίες που εκφράζονται όσον αφορά την επάρκεια του δημοσίου ελέγχου και τη διαφάνεια, όλα αυτά δημιουργούν σοβαρή απειλή όσον αφορά την υποστήριξη πλευράς γενικού κοινού για τις επιχειρήσεις του ESM και θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές εκεί που πρέπει. Τέλος, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε άλλο τομέα όπου βλέπουμε παρόμοια προβλήματα όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δημόσιο έλεγχο, δηλαδή τις δαπάνες και τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων στα κράτη-μέλη. Για 17 διαδοχικά έτη το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να δώσει γνωμοδότηση τοποθέτηση όσον αφορά το εκτικό χαρακτήρα των δαπανών ε, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο δεν δείχνει ακριβώς που έγκυται τα προβλήματα και ποιες βελτιώσεις απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους. Με βάση αυτό το ιστορικό, η Ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε εδώ και αρκετά χρόνια να παρουσιάσει το πώς χρησιμοποιούνται τα υπόρρια της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην Ολλανδία σε αιτήσια δήλωση από βάση των κρατών μελών. Η ελεκτικό μα φορέα ζήτησε να δώσει δήλωση αξιοπιστία υπό τη μορφή ανεξάρτητη νομοδότηση και αυτό κάνουμε εμεί για την έκτη φορά τώρα. Μέχρι τώρα, μόνο τρία άλλα ε, κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν κάτι παρεμφερέ. Η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο στις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις, το νέο δημοσιονομικό κανονισμό αυτό το θέμα για μία ακόμη φορά έγινε κάτι επίμαχο. Το Συμβούλιο μέχρι τώρα αρνήθηκε να δεχτεί την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμπεριλάβει υποχρεωτική δήλωση των κρατών μελών όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. Και για να χειροτερήσουν τα πράγματα, το Συμβούλιο εμένει στην αντίστασή του να δημοσιοποιεί αδίποτε μορφή έκθεσης λογοδοσία που μπορεί να ε, οδηγήσει πίσω να ταυτοποιήσει συγκεκριμένο κράτο μέλο. Αν αυτές οι εξελίξεις συζήτηση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού γίνουν αποδεκτές στο τέλος, αυτό κατά την άποψή μου και την άποψη του Αντιπροέδρου μας γυρίσει πίσω το χρόνο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής διαχείρισης Ευρωπαϊκή Ενώσεω, Κάποια χρόνια πίσω θα πάμε και θα υπονομεύσει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το σωστό δημόσιο έλεγχο. Αυτό για μας το Ελεκτικό Συνέδριο τη Ολλανδία και εσεί στην Επιτροπή σα, αυτό είναι κάτι που θέλαμε να προωθήσουμε πάντα να γίνουν αυτοί Η υπηρεσία μα πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια η πρόκληση θα είναι να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε σωστή διακυβέρνηση και καλές διευθετήσεις διακυβέρνηση όσον αφορά το μέσο της χρηματοδοτικής σταθερότητας και την εφαρμογή του προπολογισμού, την εκτέλεση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Από την έποψη του εξωτερικού ελεγκτού, ο καλύτερος τρόπος να συμβάλλουμε σε αυτό είναι μέσω συντονισμένης δράσης σε δύο επίπεδα. Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος μέλος. Μόνο μέσω του συντονισμού της διαδράσεως και αμοιβαίας ε, αλυσίδας ελέγχου και λογοδοσία σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα είναι δυνατόν να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να υπάρξει κοινό σύνδεση με το κοινό. Για το ESM, δυνατότητε για συντονισμένη δράση ήδη υπάρχουν σε ευρυονική μορφή ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου των ε, Ελεγκτών. Για την εκτέλεση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω χρειάζονται περισσότερε αλλαγέ. Είναι ο δικό σα ρόλο. Θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σα. Αν έχετε ερωτήσει όσον αφορά αυτή την παρουσίαση, θα σημειώσουμε τις παρατηρήσεις και θα διαβιβάσουμε σε αρμοδίες στην υπηρεσία μας και θα σας δώσουμε γραπτός απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Φάντεμπος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πλέον ξεκάθαρο πως Τίθεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα εδώ από την Επιτροπή μας στη σημερινή ακρόαση και νομίζω ότι είναι απαραίτητο και να το συζητήσουμε και να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Αναβάλω το επόμενο σημείο μέχρι το απόγευμα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που ε, ε, συνεργαστήκατε και το δεχτήκατε. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε χρόνο γιατί είναι βασικότατο το σημείο και τώρα θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο γύρο ερωτήσεων και τοποθετήσεων. Ας ακούσουμε την εισηγήτρια, την κυρία Ιβάνοβα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις Εθνικές Ελεγκτικές Αρχές καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που συζητήσαμε, που ήρθαμε σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν μας συμβαίνει συχνά. Πρόκειται για μια σοβαρότατη ανησυχία αυτή που εξέφρασε ο Ολλανδός συνάδελφος ε, τέλος πάντων θα περάσω σε ερωτήσεις προς τον κύριο Καλντέιρα πρώτα απ' όλα στην παρουσίασή σας είπατε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υποπτία σαν να ήταν θεσμικό όργανο από το ελεγκτικό συνέδριο και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης που υιοθετήσαμε πέρυσι. Λέμε ότι ε, ως προς τις ε, καταθέσεις των κρατών ε, που εκφράζονται σε ευρώ, αν υπάρχει θέμα αποπληρωμής μάλλον αν θα υπάρχει θέμα επιτοκίων τότε δηλαδή μια νέα πηγή εισοδήματο ε, τότε θα αρχίσει να ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός. Μήπως ε, ε, επ' αυτού θα μπορούσε να ασκήσει τον ελεκτικό του ρόλο το ελεκτικό συνέδριο. Αυτά τα έσοδα από, τα, από τους τόκους θα μπορεί να τα ελέγχει. Επίσης, ε, μπορεί να κάνει αναθεώρηση του ισοζυγίου πληρωμών ε, για το 2012 και το έχει αρχίσει να το κάνει αυτό το ελεγκτικό συνέδριο. Χαίρομαι ιδιαίτερο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, προτίθεται να κάνει άλλους τέτοιους ελέγχους, π.χ. έλεγχο του EFSM προς τις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε το άρθρο 32 εδάφιο 8 όπου λέει στο μέτρο που είναι αυτό απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων προβλέπονται στη συνθήκη όλα τα στοιχεία ενεργητικό του ESM δεν θα υπάγονται σε οδήποτε περιορισμό, έλεγχο κτλ. Δηλαδή πλήρης ασυλία. Έτσι μου φαίνεται εμένα όταν διαβάζω το άρθρο. Αυτά όμως αναφέρονται ή μάλλον αν και αντιπαραβάλλουμε τώρα τη δήλωση ε, της ε, όπου λέμε ότι οποιασδήποτε ε, συναλλαγές ασχέτως με τον τρόπο με τον οποίο καταλογίζονται στον προϋπολογισμό θα αποτελούν αντικείμενο ελέγχου για τις εθνικές ελεγκτικές ε, αρχές. Αυτό ισχύει για όλες τις διεθνείς ε, οντο, νομικές οντότητες και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει καν αυτό το άρθρο 32 εδάφιο 8 που εξαιρείται το ESM από οποιοδήποτε έλεγχο. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιβάνοβα και πριν ακούσουμε τις ερωτήσεις ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούτη που ε, μετήχε ενεργά ε, στην σημερινή ακρόαση. Ξέρω ότι έχετε άλλες υποχρεώσεις. Ε, σας ευχαριστούμε και πάλι και ευελπιστούμε να σας δούμε σύντομα στην Επιτροπή μας. Η πρώτη ερώτηση απευθυνόταν προς τον πρόεδρο Καλντέιρα, τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα μπορούσατε ίσως να τοποθετηθείτε για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις της κυρίας Ιβάνοβα. Ε, θα αρχίσω από το ευκολότερο, από το τελευταίο σημείο ε, στο πρόγραμμα εργασίας μας για το 2012 προβλέπεται έλεγχος για το ισοζύγιο πληρωμών και για το EFSM. Οι συναλλαγές σε βάση του μηχανισμού ισοζυγίου πληρωμών αρχίσαν το 2008 ε, και βλέπουμε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάληψη υποχρεώσεων και για κράτη που δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη. Όλες οι δανειοδοτικές και δανειοληπτικές δραστηριότητες πέρα από τις εγγύσεις, αλλά αυτό δεν είναι καινούριο, ε, υπάρχονται σε αυτή την ε, διάταξη. Για το EFSM, ε, άρχισαν αυτές οι δραστηριότητες το 2011 και θα δούμε τι θα μας δείξουν οι αιτήσιοι λογαριασμοί. Ε, ε, πρόθεσμα λάβαμε τους προσωρινούς λογαριασμούς, θα κάνουμε τον ελεγχό μας ε, και ε, θα σας ενημερώσουμε για αυτό το σημείο. Για τα μελλοντικά μας προγράμματα εργασίας, είναι προφανές ότι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα αιτήματα προς το δικαστήριο για τα ζητήματα προτεραιότητας. Για το 2012 έχουμε ορίσει τις ε, προτεραιότητες μας. Δεν θα ολοκληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι προσπάθειες μέσα στο 2012, αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, οι εγγύσεις του EFSF θα παραταθούν. Άρα δεν μπορούμε Ε, να περιοριστούμε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το Μνημόνιο Συνεννόησης. Νομίζω όμως ότι αυτό το είπαμε και ε, προηγουμένως. Ε, σε σχέση τώρα με την εποπτεία του ESM, εννοούσα το εξή. Το ελεγκτικό συνέδριο, καθότι είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, δεν έχει εντολή ελέγχου για το ESM. Αυτό καθ' αυτό. Απλά και μόνο διότι είναι μια διακρατική, ε, ένας διακρατικός θεσμός που εκπίπτει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπα όμως ξεκάθαρα επίσης ότι... Ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, συμμετέχουν στην εκταμίευση των δανείων από το ESM, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό προβλέπεται στη συνθήκη σύστασης του ESM. Άρα εμέσως υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσε να θεωρήσει το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα μπορούσε να εποπτεύσει, αν συντρέξει λόγος αν το κρίνουμε σκόπιμο. Σε σχέση τώρα με τον έλεγχο του νέου εισοδήματο από τους τόκους, για να επανέλθω στον προπολογισμό της Ένωσης, ε, θα δούμε πώς θα καταγραφεί στους ετήσιους λογαριασμούς. Να ξέρετε, αυτό το νέο εισόδημα δεν ε, είναι δεδουλευμένη τόκη και στη, θα μπει, θα καταλογιστεί στους ιδίους πόρους του ESM και ουχή στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η έκθεση... Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα μεριμνά ούτω ώστε οι λογαριασμοί που θα έχουν ελεγχθεί από εξωτερικό ελεγκτή θα αποτυπώνουν πίστα τα ποσά που ε, το νέο εισόδημα από τους τόκους. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι ανοίγουμε παραθυράκια, πόρτες κτλ. Απλώς λέω ότι τα ποσά που καταλογίζονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης στη συνέχεια καταλογίζονται στους ιδίους πόρους του. Ιεσέμονται δουλευμένα και θα ε, το Διοικητικό Συμβούλιο, του ESM θα μερίμνα ώστε μετά τον εξωτερικό έλεγχο να αποτυπώνουν στου αιτήσιου λογαριασμού σωστά αυτά τα ποσά. Σα ευχαριστούμε κύριε Καλντέρα. Ε, τώρα η επόμενη ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, ήταν για τον κύριο Ερμπ ε, από το Γερμανικό Ελεγκτικό. Ναι, ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα που μου απευθύνατε. Στο άρθρο 32 δεν ε, βλέπουμε να ζημιώνεται, να παρομεύεται η ελεγκτική εντολή του Συμβουλίου. Το άρθρο 32 λέει ότι ρυθμίζεται το καθεστώς ε, βάση του ελεγκτικού συνεδρίου βάσει της νομοθεσίας της ε, χώρας που έχει την έδρα του και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για την διενέργεια του ελέγχου. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ευρύ δικαίωμα πρόσβασης. Άρα λοιπόν μπορεί το ελεγκτικό συνέδριο να πετύχει κάποια έγγραφα και ε, είναι απαραίτητο να τα λάβει ούτως ώστε να διενεργήσει σωστά τον, τον απαιτούμενο έλεγχο. Κύριε Βάντε Πόστο, θέλετε να απαντήσετε όχι. Τότε θα έχουμε έναν γύρο ε, ερωτήσεων και απαντήσεων. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ο κύριο Σέντλαργκάρντ θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα προ τον κύριο Καλντέιρα. Ακούσαμε τον κύριο Βάντεν από το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο να μας λέει τα πράγματα με μεγάλη σαφήνεια περιέγραψε ε, τα κενά που υπάρχουν και τις δυνατότητες ε, που υπάρχουν ε, για τις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Θα ήθελα συγκεκριμένα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε εσείς βάσει της δικής σας εμπειρίας στο, Εθνικό, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να διεξαχθούν έλεγχοι για το ESM. Άλλη ερώτηση. Και την απευθύνω ε, στο Ολλανδικό και Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο. διαβλέπω μία μεγάλη διαφορά ως προς τις τοποθετήσεις σας και τους στόχους σας. Είναι θέμα ε, ταμπεραμέντου, είναι θέμα ε, διαφορετικής ε, τοποθέτησης, διαφορετικής άποψης. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Για ποιο λόγο δηλαδή προκρίνεται διαφορετικές προσεγγίσεις στον Πάρτιο. Έγινε μία σύσκεψη για τους εκπροσώπους των εθνικών ελεκτικών ε, συνεδρίων που εμπλέκονται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας ενημερώσετε για τις συζητήσεις ε, ε, που έγιναν. Αλλά πάντως θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα σύγκληση ανάμεσα στο Ολλανδικό και το Εθνικό Ελεκτικό Συνέδριο. Σας ευχαριστούμε. Ο Ρούμπικ τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι για μας είναι πολύ σημαντικός ο ο σχεδιασμός για το μέλλον να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Γιατί μέχρι το 2020 θα ήταν δυνατό για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να, να καταλήξει ένα είδος scoreboard, ένα πίνακα αξιολόγηση για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τα τρία αυτά εργαλεία ε, πώς εξελίσσονται οι αριθμοί, τι γίνεται με τις επιστώσεις, με τις εγγύησει και το διοικητικό κόστος. Νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να έχουμε μια τέτοια εικόνα ε, να έχουμε αυτούς τους αριθμούς ε, τη ίσως εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Να δούμε κατά πόσο τηρούνται ε, οι προγραμματισμοί, ε, τηρείται το πρόγραμμα και ή όχι. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό πλαίσιο, ε, κάνουμε προγραμματισμό με το 2020. Τι θα συνέβαινε εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτά τα 60 δις που προβλέπει το χρηματοπιστωτικό πλαίσιο ε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τι θα συνέβαινε εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρνεί να δώσει τη συγκατάθεσή του. Επίσης ε, προς το γερμανό ε, εκπρόσωπο του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τον ε, εθνικό προγραμματισμό του, για τον προγραμματισμό μάλλον του εθνικού προπολογισμού. Ε, έχετε συγκεκριμένους αριθμούς, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Έχετε επίσης μια εικόνα εν σχέση με το ποιες θα είναι οι συνέπειες και επιπτώσεις μέχρι το 2020. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούμπιχ. Δίνω το λόγο στον άλλο κύριο Ουντή. Δύο παρατηρήσεις. Ε, πρώτον, σε σχέση με τον ε, τεχνικό έλεγχο, δεν κατάλαβα καλά. Όταν μιλούσατε για το άρθρο 30, ε, ε, η, αυτή η Επιτροπή των Ελεγκτών είναι πέντε συν τρία μέλη ή πέντε εκ των οποίων τα τρία. Γιατί δεν είναι σαφής η διατύπωση. Ε, ε απαρτίζεται από πέντε μέλη η Επιτροπή και λέμε ότι διορίζονται κάποια μέλη βάσει προτάσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν, δεν είναι ξεκάθαρο για μένα αν είναι τρία από τα πέντε μέλη. Τέλο πάντων, για τον τεχνικό έλεγχο νομίζω ότι την πατήσαμε όλοι. Γιατί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρότειναν και να ε, επενέσω επ' αυτού και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Μας, ε, εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να συμπαραταχθεί. Λοιπόν, για αυτήν την ελεγκτική επιτροπή. Ποια μέσα θα έχει στη διάθεσή της για να επιτελέσει την αποστολή της, θα έχετε συνεργάτες, σε ποιο προϋπολογισμό, τι προϋπολογισμό θα έχετε στη διάθεσή σας. Δεύτερον, όταν ε, όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 σχετικά με τους ανεξάρτητους ελεγκτές, ε, ε λοιπόν με ξαφνιάζει ότι η παρουσία εξωτερικών ελεγκτών δεν προβλέπεται για την, εσωτερική ελεγκτική επιτροπή. Εγώ θα θεωρούσα φυσιολογικό ε, τουλάχιστον ε, η εσωτερική ελεγκτική επιτροπή να ακούει τις γνωμοδοτήσεις των εξωτερικών ελεγκτών. Η ανεξαρτησία λοιπόν των εξωτερικών ε, ε, ελεγκτών στο άρθρο 29 δεν μπορεί να διαφυλαχθεί μέσω της απαγόρευσης αποστολών επιτόπου στα κράτη-μέλη ενώ αυτό θα προαγάγει την ε, αίσια λειτουργία του ολόκληρου του μηχανισμού. Άλλο που με προβληματίζει είναι ότι δεν υπάρχει τραπεζικός κανονισμός. Μιλάμε για έλεγχο των ετησίων λογαριασμών, δεν μιλάμε όμως για σύσταση πιστοτικών ιδρυμάτων και τον έλεγχο αυτόν διότι στον κόσμο των οικονομικών αυτό θα ε, παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο. Ε, σας συγχαίρω διότι επεκτείνατε την εντελή στη διαχείριση, προτείνατε να επεκταθεί η εντολή σα στη διαχείριση ε, των κινδύνων. Ελπίζω να το πετύχετε, αλλά ξέρετε μία απλή δραστηριότητα εξωτερικού οικονομικού ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα γενικότερο πλαίσιο για τι τραπεζικέ συναλλαγέ και δεν έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα είναι ο έλεγχος των λογαριασμών. Το πρόβλημα είναι ο πολιτικός έλεγχος ε, και ε, πού είναι αυτός ο πολιτικός έλεγχος για ε, τα τόσο υψηλά σημαντικά κονδύλια. Δεν υπάρχει καν διαδικασία απαλλαγής. Δηλαδή τα μέλη της κυβέρνησης αυτοχορηγούν χορηγούν στον εαυτό τους την απαλλαγή για την εκτέλεση των προϋπολογισμών αυτών των νέων οργάνων και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεν δέχτηκαν τον πολιτικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι δημοκρατική αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει προηγούμενο. Ελπίζω να διορθωθεί η κατάσταση είναι άγωνη αυτή η διάκριση που γίνεται ανάμεσα στο διακρατικό και τον ε, ενωσιακό χαρακτήρα κάποιων θεσμικών οργάνων νομίζω πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και τουλάχιστον για τους μόνιμους μηχανισμούς σε οποιοδήποτε δημοκρατικό πολίτευμα όταν υπάρχει χρήση δημοσίου χρήματος και το είπατε κι εσείς ε, κύριε ότι προβλέπετε έλεγχος από ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Ε, λοιπόν, σε οποιοδήποτε τέτοιο πολίτευμα προβλέπεται ε, πολιτικός έλεγχος βάσει λαϊκής εντολής. Εδώ δεν προβλέπεται. Για την απαλλαγή για τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να θυμόμαστε ότι καλύπτονται 17 κράτη από αυτό το μηχανισμό και δεν υπάρχει καμία κοινοβουλευτική διάσταση. Δηλαδή προσπαθούμε να οικοδομήσουμε οικονομική διακυβέρνηση βάσει όμως αρχής διακρατικότητας ε, των κυρώσεων και ό,τι θέλετε αλλά ε, χωλαίνει ε, ε, το όλο εγχείρημα διότι δεν έχουμε αυτή την, κοινοβουλευτική διάσταση. Πώς θα καταφέρουμε να έχουμε δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό πολιτικό έλεγχο σε αυτό το υποσύνολο εφόσον ε, επιθυμούμε να οικοδομήσουμε οικονομική διακυβέρνηση, να έχουμε όργανα που εξασφαλίζουν σταθερότητα και να διαφυλάξουμε το νόμισμα. Ε, ε, Ευχαριστούμε κύριε Όντι. Αναφερθήκατε σε ένα σημαντικό θέμα. Πρόκειται για ποσά τα οποία αποτελούν το πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να θέτουμε εδώ το ερώτημα σε σχέση με τον έλεγχο, δηλαδή ποιος ελέγχει τη χρήση αυτών των χρημάτων, ε, ποιες παράμετροι επιλέγονται. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να απευθύνω προς τον κύριο Έρ. Πώς αξιολογεί εκείνος το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, δηλαδή τη ενέργειες ελέγχου εκ μέρου των Εθνικών Κοινοβουλίων και βεβαίως εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα ήταν το δικό μου ερώτημα το οποίο θα ήθελα να εκφράσω υποστηρίζοντας την παρέμβαση του κυρίου Οντί. Έχουμε επίσης τον κύριο Μούλτερ που θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Μούλτερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ζήσα το λόγο. Θα υπογραμμίσω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Οντί. Νομίζω ότι είμαστε στο μονοπάτι το διακυβερνητικό άνευ κοινοβουλευτικού ελέγχου και αυτό αντιβαίνει τις εξελίξεις της τελευταίας 20 ετίας, 30 ετίας και ε, περνάμε δύσκολες περιόδους στην οικονομία μεν, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τη στην Ευρώπη χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ξεκινάμε έναν δρόμο που είναι πολύ επικίνδυνος κατά την άποψή μου και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Οντί. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στους συναδέλφους των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων για τελευταίο σχόλιο που θα απευθύνουν προς τον ε, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και για τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν εδώ. Ίσως ε, θα, θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Δηλαδή, κατά πόσο υπάρχει μια διαφορετική σκοπιά ε, στο θέμα του εξωτερικού ελέγχου μεταξύ δηλαδή Γερμανών και Ολλανδών συναδέλφων. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το οποίο παρουσίασα εγώ εδώ αντανακλούν τις ε, θέσεις ε, τις οποίες εκφράζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και έχει συμφωνήσει με το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο το Μάρτιο του περασμένου έτους και ε, στις οποίες συμμετείχαν επίσης και συνάδελφοι από άλλα ελεγκτικά συνέδρια και από το Ολλανδικό και κατέληξαν σε μια συμφωνία. Συνεπώς ε, τα όσα είπα εδώ τελικά αντανακλούν μια κοινή αξιολόγηση και κοινέ προτάσεις για μια ρύθμιση του εξωτερικού ε, ελέγχου και έτσι όπως θα πρέπει να εδρεωθεί στη συνθήκη καθώς και τις προτάσεις που θα έπρεπε να περιληφθούν στο καταστατικό. Ασφαλώς ε, υπάρχουν κάποια σημεία τομείς βρέθηκε ένα σκληρό παρανομαστή όσον αφορά τι διάφορε προσεγγίσει. Το Μάρτιο στη Βόνη συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα ε, σε ποιο βαθμό το Board of Auditors, το ελεγκτικό συμβούλιο, μπορεί να εξετάσει τα προγράμματα και την οικονομική αποδοτικότητα. Και τελικά ε, συμφωνήσαμε να αποδεχτούμε τη διατύπωση ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους των προγραμμάτων. Τώρα, σε ποιο βαθμό οι έλεγχοι αυτοί ε, υπερβαίνουν τα όρια που είχε θέσει το, το Συμβούλιο Διακυβέρνησης για τα βοηθητικά μέτρα. Δηλαδή κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει μια εντολή για, μια εξωτερική, για ένα εξωτερικό έλεγχο του FSM. Ε, αυτό δεν έχει οριστικά το Μάρτιο. Και βεβαίω υπάρχουν εδώ διαφορετικές απόψεις. Και θεωρώ ότι ο Ολλανδό συνάδελφος σε αυτό αναφέρθηκε εδώ. Ε, θα πρέπει, ωστόσο, έστω και αν έχουν γίνει, όπως σας είπα, σχετικοί προβληματισμοί, θα πρέπει να τονίσει κανείς και θα πρέπει να αναγνωρίσει και νομίζω ότι τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια μπορούν να είναι ιδιαίτερα περήφανα γι' αυτό, ότι από τη δική μας σκοπιά, από τη γερμανική σκοπιά, ε, έχει υπάρξει μία συμφωνία όσον αφορά σημαντικά θέματα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένας εξωτερικός έλεγχος και να διατυπώνεται αυτό στη συνθήκη και να συμφωνεί με τις διεθνείς προδιαγραφές. Σε ποιο βαθμό τώρα υπάρχουν πολιτικές ανάγκες ε, διεξαγωγή ελέγχου εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων και των Εθνικών Κοινοβουλίων, αυτό μπορώ να το κατανοήσω, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω. Από εθνική σκοπιά το Bundesrechnungshof, το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει, ε, μάλλον να ελέγχει τις ε, οικονομικές ε, δραστηριότητες. Αλλά βεβαίως, δηλαδή του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, βεβαίως εδώ προσκρούει κανείς τα όρια των πολιτικών αποφάσεων και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη του εξετάζοντα την πολιτική κατάσταση καταρχήν από γερμανική σκοπιά και θα πρέπει βεβαίω και να το σεβαστεί, τουλάχιστον έτσι όπω εμφανίζεται από τη δική μα πλευρά. Όσον αφορά τώρα τι ε, επιπτώσει στο γερμανικό προπολογισμό, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, υπάρχουν μια σειρά από νομοθετικά, νομοθετικές δέσμες, πακέτα μεταξύ αυτών για έναν διορθωτικό προϋπολογισμό ο οποίος ε, είναι αναγκαίος ε, σε σχέση με τις ε, πληρωμές ρευστό στο ESM μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε έναν μεσοπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό στη Γερμανία μέχρι το 2015 και στο πλαίσιο αυτό ε, προβλέπονται αυτές οι προκαταβολές. Η μεσοπρόθεσμος ε, οικονομικός προγραμματισμός έχει μια ενημερωτική λειτουργία για το Κοινοβούλιο, δεν είναι δηλαδή δεσμευτικός, αλλά στο βαθμό που προβλέπονται κάποιες πληρωμές από τον τρέχοντα και από τον επόμενο προπολογισμό όσον αφορά αυτά τα 18 δις, γιατί η Γερμανία θα πρέπει να καλύψει το 27%. Ε, αυτά, όπως σας είπα, λαμβάνονται υπόψη στον διορθωτικό προπολογισμό και στον προπολογισμό του επομένου έτους. Ε, στη Γερμανία έχουμε ε, ένα συνοδευτικό πακέτο για τη διακυβέρνηση ε, ένα, μια φορολογική δέσμη, ένα φρένο, μια τροχοπέδη για το χρέος, το οποίο από το 2020 ε, προβλέπει ένα έλλειμμα της τάξης του 0,35% ε, ε, μετά το 20% για όλους. Τώρα, για να αντιμετωπίσω το θέμα του χρέους στη Γερμανία, έχουμε ένα 80% του ΑΕΠ, από το 2013 γιατί μπήκαν και στο πρόγραμμα σταθεροποίησης από το 2015 θα μειώσουμε το επίπεδο του χρέους από το 80% στο 60%. Και εδώ γίνεται μια διεξοδική συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και κρατηδίων. Δεν έχουμε καταλήξει. Τώρα όσον αφορά το ελεγκτικό συμβούλιο των τριών ή πέντε μελών, όπως αναφέρθηκε εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε ως εξή. Οι τρει βεβαίω είναι ε, τμήμα των πέντε, δηλαδή συνολικά έχουμε πέντε μέλη, τρία από αυτά θα είναι εκπρόσωποι ελεγκτικών συνεδρίων, ε, θα υπάρχει και ένα εξ αυτών ένας θα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο άλλοι θα διορίζονται εκ περιτροπή από εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια αναλλαγή μεταξύ των δικών μα αντιλήψεων, δηλαδή ε, χωρών που έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στο ESM και χωρών που έχουν ένα μικρότερο μερτικό στο ESM. Ωραία λοιπόν. Ε, και το εναπομείναν ερώτημα από τον πρόεδρο ε, προσπάθησε να το απαντήσω το ερώτημα του ποιος ελέγχει τις ε, αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Από τη δική μας πλευρά του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, εδώ βρισκόμαστε στο πολιτικό πεδίο. Στη Γερμανία υπάρχει μια έντονη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε σχέση ακριβώς με την αύξηση των ε, κονδυλίων καθώς και με την ε, νομοθετική εδραίωση του FFSF ε, στη Γερμανία σημαντικές αποφάσεις που δεν βρίσκονται κάτω από τεράστια ε, χρονική πίεση για την έγκριση βοηθητικών μέτρων βρίσκονται υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ε, η Γερμανία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και τόνισε την αναγκαιότητα λήψη κοινοβουλευτική απόφαση στα θέματα αυτά. Το τόνισε ρητά και εντόνως και ως εκ τούτου υπάρχει, θεωρώ, μια σημαντική κοινοβουλευτική συμμετοχή. Ε, βεβαίως, εάν τα μέτρα είναι κατεπίγουσας φύσης, ε, υπάρχει μια κάλυψη από τον νόμο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Έρπ. Ο κύριος Βάντεπούς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα εντάχει να σχολιάσω τη διαφορετική προσέγγιση που παρατηρήσαμε ανάμεσα στο Ολλανδικό και το Γερμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσετε το ερώτημα που μας θέσατε. Έχουμε κατά τη ευρύτερη προσέγγιση σε σχέση με την, το Ολλανδικό Ελεγκτικό Συνέδριο. Βεβαίως, όπως και εκείνη, δηλώνουμε ικανοποιημένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και την πρωτοβουλία κυρίως των Γερμανών συναδέλφων μας υπό την αιγίδα του Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την συζήτηση των ελεγκτικών διατάξεων ε, και του ESM. Είναι πολύ καλές συζητήσεις που γίνονται για αυτά τα δύο ζητήματα. Στην παρουσίαση ο Γερμανός συνάδελφος τόνισε παρκώς αυτά τα θέματα. Τώρα από πλευράς μας προσεγγίσαμε το θέμα της ακρόασης λίγο διαφορετικά. Για μας η καλή διακυβέρνηση είναι αναπόσπαστο τμήμα της σωστής στρατηγικής εφόσον μιλάμε για ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή και εστιάζουμε στις τρεις βασικές αρχές, δηλαδή διαφάνεια, λογοδοσία και δημόσιος έλεγχος. Ο αντιπρόεδρος μας ε, εξέτασε ε, τι γίνεται σε μια, μια ιδανική κατάσταση και στην πράξη αυτά ε, κάνουμε και γι' αυτό ακουστήκαμε πιο επικριτική από ό,τι οι Γερμανοί συνάδελφοι παρόλα αυτά συμφωνούμε μαζί τους ότι έχουν ήδη γίνει πάρα πολλά και συνεχίζουν ε, να βελτιώνται τα πράγματα ως προς την διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Καλντέιρα τώρα. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαι σύντομος γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θα δώσω ταχύτατες ε, απαντήσεις. σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Σέντεργκάρντε... το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνεδρίο έχει ξεκάθαρη εντολή να ελέγχει δηλαδή τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι διεθνείς οργανισμούς Συμφωνήσαμε με τις εθνικές ελεγκτικές αρχές ότι υπάρχει ένα κενό ως προς, ε, τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο. Ε, όπως σωστά ανέφερε και ο κύριος Σοντή και αυτό σχετίζεται με τις νέες εξελίξεις ε, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ε, κυρίως ε, ως προς τα κράτη της Ευρωζώνης. Αυτά λοιπόν που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ε, ταιριάζει με μία απάντηση στο βαθμό του δυνατού, σε μία ανταπόκριση με το έλλειμμα του δημόσιου ελέγχου και τη λογοδοσία όσον αφορά το EFSF και με διάφορες διευθετήσεις που αφορούν το ESM που όπως αναφέρθηκε ίσως θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα του δημοσίου ελέγχου από πλευρά ε, κοινοβουλίων όσον αφορά τη λογοδοσία. Υπάρχουν ε, θέματα διαφάνειας, υποβολή αναφορών στα εθνικά κοινοβούλια, αφού πήγαμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη κυβερνητικό πεδίο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει πώς μπορεί να διευρύνει περαιτέρω τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια όπως και με τα άλλα εθνικά, με εθνικούς φορείς. Κύριος Ρούμπινγκ. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επιθυμεί διακαώς να κάνει τα δέοντα, όχι μόνο όσον αφορά τη χρήση των χρηματοδοτικών αυτών μέσων, αλλά εν γέννη. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουν, πώ να το πω, εκθέσει τοπίων του ΣΥΠΗ, γενική εικόνα. Θα την προωθήσω αυτή την ιδέα. Και όπως κάναμε και με γνωμοδότηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημοσιεύθηκε το 2010, και εδώ, και εδώ, με αυτό το εργαλείο θα πρέπει να παρέχουμε γενική επισκόπηση των χρηματοστατικών μέσων που χρησιμοποιούνται για αυτή την οικονομική και χρηματοσυντική κρίση. Υπάρχει μακράς διαρκείας ευθύνη ανάλογα με την οριμότητα των δανείων και αυτό θα πρέπει να παρακολουθείτε δεόντως όσον αφορά το EFSM και οι υποχρεώσεις όσον αφορά τα 60 δις του EFSM ε, και αυτές οι υποχρεώσεις θα πρέπει να τηρηθούν. Και εδώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να έρθω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέγε Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλδέρα. Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα για να συνοψίσει και επίσης να κάνει κάποιες ε, προτάσεις για την ε, συνέχεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμμετέχοντες σε αυτή την κρόαση γιατί πραγματικά με τις παρατηρήσεις τους έδωσαν τη βάση για μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, Ζανκάλ, κύριε Άνεφ, ε, καθώς και τον κύριο Μπούτι, ο οποίος έπρεπε να, εγκαταλ... μας εγκαταλείψει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αλλά και τους εκπροσώπους των Εθνικών ελεκτικών Οργάνων, τον κύριο Έρπ και τον κύριο Βάντεμπρος, αλλά ιδίως, και εσάς κύριε Καλδέρα. Πραγματικά ε, σχηματίσαμε την εντύπωση ότι ασχολείστε ο ίδιος εντόνως με αυτό το θέμα της υποχρέωσης λογοδεσίας και της διενέργειας ελέγχων αλλά νομίζω και μπορώ να το συνοψίσω από τη δική μου πλευρά ότι μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις, μάλλον χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις για να διευκρινιστούν τα θέματα τα οποία εκκρεμούν ακόμα. Ε, σημαντικά θέματα όσον αφορά το μεγάλο όγκο των χρημάτων. Σε αυτό άλλωστε αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί εδώ θα πρέπει να κλείσουμε ε, αυτό το χάσμα, το έλλειμμα του δημοσίου ελέγχου, γιατί το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος. Και γι' αυτό ε, πραγματικά είμαι ευγνώμων ε, προς την κυρία Αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας, την κυρία Ιβάνοβα, η οποία έχει προωθήσει τόσο πολύ, τόσο ενεργητικά το ζήτημα αυτό. Και θα ήθελα να της δώσω τον ε, τελικό, του καταληκτήριο λόγο Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τους ειδικού και δίνω το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την ε, πολύ χρήσιμη συζήτηση που μπήκε σε μεγάλο βάθος. Ευχαριστώ και τους ε, αγορητές, ομιλητές μάλλον. Τα βασικά ερωτήματα των συναδέλφων αναφερόταν σε κάποια θέματα όπως ε, η χρήση του EFSM σε σύγκριση με το EFSF ή ESM, ε, ποια είναι η τάση, θα αλλάξει, θέματα που αφορούν τη συνύπαρξη του EFSF με το ESM και ποια θα είναι η διαδοχή των δύο προσωρινών μέσων με το μόνιμο μέσο και ο Σμόλτερ αναφέρθηκε επανειλημμένο στο δικαίωμα ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το ESM. το θέμα. Ο κ. Γκάιερ αναφέρθηκε στο θέμα του κόστους διαχείρισης, ποιο θα είναι. Ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ήταν τόσο αισιόδοξη όσον αφορά τις αποπληρωμές ε, και εγώ συμμερίζομαι την άποψη σου και Σοντή αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το δημόσιο έλεγχο και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, υποστηρίζω τον κύριο Ρούμπικ στο αίτημά του για ένα σύστημα βαθμολόγησης scoreboard και χαίρομαι ότι ο κύριος Καλτέρα θα υποβάλει σχετική πρόταση για την υποβολή αυτή της επισκόπησης, της έκθεσης που θα δίνει μια γενική εικόνα. Συνοψίζοντας, θέλω να στείλω τέσσερα μηνύματα που διαμορφώθηκα μετά τη συζήτηση κατά την άποψή μου. Δεν αφισβητούμε την χρησιμότητα αυτών των χρηματοσφικών μέσων. Χρειάζονται κατεπηγόντως. Είναι ζωτική σημασία για να διασωθούν κάποια κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτό που αμφισβητούμε είναι η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και ο έλεγχο αυτών των μέσων και οι φορολογούμενοι τη Ευρωπαϊκή Ενώση έχουν δικαίωμα να ξέρουν ποια είναι τα αποτελέσματα και πώ χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα. Χρησιμοποιήθηκαν σωστά και το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει αυτό το δημοκρατικό έλεγχο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, έχουμε 110 δισεκατομμύρια ευρώ ε, υποχρεώσεις όσον αφορά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και χρωστάμε στους πολίτες ε, τον ε, δημόσιο έλεγχο, τον δημοκρατικό έλεγχο των ευθυνών που έχουν αναλυφθεί και των υποχρεώσεων. Καλωσορίζω μετά την πρόθεση που εκφράστηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο να ξεκινήσει η ανάλυση του συζυγίου πληρωμών φέτος και ελπίζω ότι αυτό το βήμα θα ακολουθηθεί με την έκθεση τοπίου, τη γενική επισκόπηση και την περαιτέρω ανάλυση των χρησιμοποιητικών εργαλείων. Και τέταρτον και σημαντικότερο, καλούμε και θα καλούμε συνεχώς να παίξει μεγαλύτερο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με όλες τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν από το FSM μέχρι τη ε, διαδικασία του προπολογισμού, απαλλαγή, ESM. Είναι υποχρεωτικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απορρέουν από τις εκθέσεις για το ESM, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα εθνικά. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζητούμε κατ' μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία και στη διαδικασία της αναπτύξεως του εσωτερικού κανονισμού που θα διέπει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση. Ο πολιτικό έλεγχο είναι βασική μα προτεραιότητα και νομίζω ότι αυτή η ακρόαση θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή περαιτέρω δράσεων θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου όλου του ομιλητέ, όλου του συναδέλφου για τη συνεισφορά του και προσβλέπω σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ.